Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και χαίρομαι που βλέπω και πολλούς ε, παρόντες τόσο νωρίς. Εγώ δυσκολεύτηκα να σκόφω γιατί όπως και εσείς ε, είχα κάποιες χριστουγεννιάτικες υποχρεώσεις, κάποιες εκδηλώσεις να παρευρεθώ χθε. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε μια συμφωνία για τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα. Χαίρομαι που η κυρία, Τάιλερ, η κυρία Στάιλερ μάλλον, είναι ακόμα εδώ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Στάιλερ να ενημερώσετε την ομάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την δυνατότητα. Την ε, Τρίτη το απόγευμα είχαμε μία σχεδόν τριών ωρών και ενός τετάρτου και καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Νομίζω ότι υπήρξε και σχετική συμφωνία στην Κορεπέρ χθε μεσημέρι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τώρα έχουμε ένα πακέτο για το Γενάρη που θα πρέπει να ψηφίσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραμε να γίνουν δεκτά πολλά από αυτά τα οποία εμείς υποστηρίζαμε στην Επιτροπή μας. Φυσικά και εμείς κάναμε κάποιους συμβιβασμούς τεχνικού χαρακτήρα ορισμένοι συμβιβασμοί και κάποιοι άλλοι συμβιβασμοί αλλά γενικά είναι ενδιαφέρον γιατί το Συμβούλιο ε, άρχισε να εννοώ. Πιστεύω ότι μας δίνει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία περίμενε κανείς. Πάντως υπήρξε συνεργασία πάρα πολύ καλή και μεταξύ των συναδέλφων και με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Πάρα πολύ παραγωγική συνεργασία και χαίρομαι που επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Μάλκομ γιατί προείδρευσε κατά πάρα πολύ ωραία τις διαπραγματεύσεις και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ για τη σκληρή δουλειά. Αν λάβει κανείς υπόψη και τις τροπολογίες που είχαμε στη δεύτερη ανάγνωση, δεν ήταν και τόσο εύκολο νομίζω να συμφωνήσει και το Συμβούλιο για τις ε, τροπολογίες της δικής μας Επιτροπής. Ευχαριστώ λοιπόν. Φαντάζομαι το Γενάρη πριν, πριν ψηφίσουμε στην Ολομέλεια θα μπορείς να μας παρουσιάσεις περισσότερα αναλυτικά τα πράγματα αυτά. Θέλω να σας πω ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η σημερινή μας συνεδρίαση, όπως νομίζω όλες οι συνεδριάσεις μας, ένα πρόσθετο σημείο για όσους βλέπουν από το διαδίκτυο την συνεδρίασή μας. Θα σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνω κάποιες ε, προτάσεις για το πώς θα βελτιωθεί η παρουσίαση των εργασιών. Θα σας διαβιβάσω ή αργότερα σήμερα τη ε, διάρκεια της εβδομάδας τις ιδέες μου για να ακούσω και τα δικά σας σχόλια. Θα θέλαμε επίσης να υπάρχει ένα σύστημα καταλόγου κατά κάποιο τρόπο, index, ε, που να μπορούν κάποιοι να αναφέρονται, να μπορούν να βρουν πιο ε, μετά τις ε, εργασίες μας στο διαδίκτυο. και θα μπορούσατε αν είχατε κάποιες ειδικέ κάρτες να προσθέτετε το όνομά σας στο, στο transcript της μετάδοσης. Έχετε λοιπόν τις κάρτες, μπορούμε να τις δοκιμάσουμε σήμερα. Αυτό έχει να κάνει και με τη γενικότερη εργασία που κάνουμε για να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας προς τα έξω. Είχα κάτι αναφέρει τελευταία φορά νομίζω, δηλαδή ότι το newsletter, το ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής μας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Όποιοι θέλετε να εγγραφείτε στο διαδίκτυο μπορείτε να το κάνετε. Έχουμε φτάσει στους χίλιους συνδρομητές ήδη και αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρει η δουλειά μας. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν, όσους μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο τόσο νωρίς το πρωί. Περνάμε τώρα λοιπόν σε έναν γύρο ακόμη της ε, συζήτησης της έκθεσης του Αντρέα Σφαπ για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έχουμε δύο ενημερωτικά έγγραφα που θα παρουσιάσουμε και οι θα κάνουν τα σχόλιά τους. Χαίρομαι για την παρουσία του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Γνωρίζω ότι υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στο Συμβούλιο στην Κορυπέρ συγκεκριμένα στο τέλος Βιλκής Προεδρίας όπου εγκρίθηκε χθε η πρόταση και φαντάζομαι ότι ε, και ο εισηγητής μας θα θέλει να μας πει κάποια πράγματα. Θέλετε να μιλήσετε τώρα, μετά από την Κομισιόν και το Συμβούλιο, εσείς θα μου πείτε. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, βέβαια, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη συνάδελφο κυρία Στάιλερ για τη δική τη την επιτυχημένη δουλειά και ελπίζω μετά από κάποιε εβδομάδε ε, να μπορώ να πω ότι με τη βοήθεια του Προέδρου ε, και χάρη τη παρουσία του θα καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή η οδηγία και να κάνει παραχωρήσει στο Συμβούλιο. Αυτή η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από δύο βασικά γεγονότα όσον αφορά την οδηγία. Εκτό από αυτά τα ενημερωτικά σημειώματα, τα briefing notes, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, αλλά καταρχήν θα ήθελα να παραπέμψω στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το Alpenhof. Ε, πριν από ένα χρόνο αναφέρθηκα σε αυτό. Αυτή η απόφαση Alpenhof αναφέρει τα εξή. Ε, ένα Αυστριακό ε, ε, είχε κλείσει ένα δωμάτιο σε αυτό το ξενοδοχείο το Alpenhof και κάποια στιγμή ακύρωσε την κράτησή του και είπε ότι η ακύρωση πρέπει να γίνει με βάση το γερμανικό δίκαιο. Γιατί ω Γερμανό προστατεύεται από το γερμανικό δίκαιο περί προστασία καταναλωτού, ακόμα και έχει κλείσει δωμάτιο στην Αυστρία. Ε, το Κοινοβούλιο έθεσε το εξή ερώτημα. Κατά πόσον αυτό το homepage της, ε, του Αυστριακού Ξενοδοχείου, κατά πόσον αυτή η ιστοσελίδα ρυθμίζεται από το γερμανικό δίκαιο ή όχι. Η ε, προστασία καταναλωτή λέει ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα εναρμόνισης γιατί έτσι κι αλλιώ ο καταναλωτή προστεύεται πάντα από το δικό του το εθνικό δίκαιο. Τώρα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Τρίτη αποφάσισε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο αλλά ότι ο Γερμανό καταναλωτή υπάγεται και ε, οφείλει να σέβεται το αυστριακό δίκαιο γιατί αυτή η αυστριακή ιστοσελίδα δεν έχει αρκετέ γλώσσες ε, και πληροφορίες για να δώσει την εντύπωση στον ε, Γερμανό καταναλωτή ότι πρόκειται για μία ιστοσελίδα που θέλει να τον προστατεύσει. Το θέμα είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν έχουν μία ιστοσελίδα στο ε, διαδίκτυο ε, δεν μπορούν να θεωρούν ότι η δική τους ιστοσελίδα λαμβάνουν υπόψη από 26 διαφορετικά κράτη-μέλη. Αλλά εκτός αυτού ε, ισχύει το ότι οι καταναλωτές οι οποίοι κάνουν δύο διασυνοριακές αγορές δεν μπορούν να θεωρούν αυτόματα ότι προστατεύονται από το δικό τους εθνικό δίκαιο περί προστασίας καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με τις προεκτάσεις αυτής της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαστηρίου στην την περίπτωση, όπω σα είπα, την περίφημη Alpenhof, ξενοδοχείο Alpenhof. Κατά δική μου άποψη είναι απόλυτο σαφέ ε, ότι η οδηγία για την προστασία καταναλωτή στην Ευρώπη, κυρίω για διασυνοριακέ αγορέ, πρέπει να ε, τύχει εναρμόνιση σε όλα τα κράτη-μέλη. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ θερμά την Βελγική Προεδρία, κυρίω τον Μίχαλ Αντενχοφ, ο οποίο με τεράστιε προσπάθειε συνέβαλε πράγματι το Συμβούλιο, το οποίο στην αρχή ήταν διχασμένο για την οδηγία, εν τέλει να συμφωνήσει και νομίζω λοιπόν ότι λόγω των διαφορετικών προϋποθέσεων που ισχύουν για την προσέγγιση δεν ε, είναι αρνητικό το να ε, πενέσουμε την Βελγική Προεδρία. Πρέπει να το πούμε. Η Βελγική Προεδρία έκανε θαυμάσια δουλειά. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι όχι μόνο γενικά αλλά και πιο ειδικά στα δύο θέματα επί των οποίων θα παρουσιαστούν σήμερα ενημερωτικά σημειώματα θα μπορεί ε, να τοποθετηθεί ε, αποτελεσματικά. Το θέμα είναι ότι η οδηγία αυτή δεν πρέπει να αντιφάσκει με άλλε οδηγίε. Πρώτον με την οδηγία e-commerce και δεύτερον με την οδηγία περιπαροχή υπηρεσιών αλλά και γενικότερα το σύνολο του τομέα περιπαροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν όσον αφορά την ε, σχέση αυτής της οδηγίας της προστασίας του καταναλωτή με άλλες οδηγίες πρέπει και το έκανα ήδη συνέστησα, συνέταξα δύο ενημερωτικά σημειώματα τα οποία και θα σας παρουσιάσω. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την οδηγία προστασία καταναλωτή, επικαλύπτεται με τις οδηγίες e-commerce, ε, ε, Anti-Commercial Practices Directive, η υποχρέωση ενημέρωσης ε, και σε αυτό το αποτέλεσμα καταλήγουν τα, οι μελέτες, η υποχρέωση ενημέρωσης από τις δύο διαφορετικές οδηγίες που προανέφερα άλλοι συμπληρώνονται, άρα δηλαδή εδώ δεν υπάρχει αντίφαση και ως εκ τούτου δεν ε, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι ε, διαφωνίες που υπάρχουν στην οδηγία περί προστασίας του καταναλωτή. Οι δύο λοιπόν αυτές οδηγίες όπως σας είπα εν μέρει επικαλύπτονται χωρίς να είναι ταυτόσιμες. Και τέλος ε, η υποχρέωση ενημέρωσης σε άλλους οδηγίες που ισχύουν δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε άλλα κενά. Εμείς λοιπόν προτείνουμε η οδηγία περί προστασίας καταναλωτή ε, θα πρέπει να καλύπτει και να δέχεται την, ε, και να συμπληρώνει περισσότερο την υποχρέωση ενημέρωση των άλλων οδηγιών. Άρα δηλαδή οι οδηγίες μπορούν να παραμείνουν όλες παράλληλα και η ελάχιστη ενημέρωση να ξεπερνάει αυτό το οποίο προβλέπεται σήμερα στις άλλες οδηγίες. Δηλαδή η, η υποχρέωση ενημέρωση που ήδη υπάρχει παραμένει άφηκτη. Όσον αφορά την οδηγία περί παροχής υπηρεσιών, το δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα λέει ότι η σχέση ανάμεσα στην οδηγία περί του καταναλωτή και την οδηγία για τι χρηματοπιστωτικές αλλαγέ. η σχέση είναι πολύ περίπλοκη. Ναι, μεν γίνονται συγκεκριμένε προτάσει το πώ ακριβώ μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά κενά, αλλά κατά τη δική μου την άποψη ε, η οδηγία περί Παροχή υπηρεσιών σήμερα καλύτερο θα ήταν να αρθεί, τουλάχιστον το άρθρο 2 να αρθεί, γιατί αυτό ε, σημαίνει ότι μπορούμε κάπου αλλού να ρυθμίσουμε τα θέματα που θίγει αυτό το άρθρο. Και τέλος ήθελα να ευχαριστώ θερμά τους σκιώδης οι οποίοι εργάστηκαν επίσης σκληρά. Ευχαριστώ και όλους τους συναντέλφου ε, που θα λάβουν το λόγο να τοποθετηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, thank σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέας. Θα ήθελες να έχουμε πρώτα μια ανταλλαγή απόψεων με τους σκιώδεις ηγητές και μετά να μιλήσει στο Συμβούλιο. Αντικαθιστάτε, νομίζω, την κυρία Γκέμπχαρτ. Θέλετε να μιλήσετε για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Όχι, ο κύριος Ρόσφορντ είναι εδώ, του Ποιος είναι εδώ τελικά. Α, ο κύριος Μπίλε. Πάλι καλά. Um, και ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι εδώ. Λοιπόν, ποιος θέλει να μιλήσει από τους σοσιαλδημοκράτες πρώτος κάποιος. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπίλαν, νομίζω είστε ο πρώτος από τους οριστέντες και ηγητές που είστε παρόν. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας κάνουμε την τιμή, σας δώσουμε το λόγο πρώτο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την πλευρά μου, θα ήθελα, συγγνώμη υπάρχει ένα πρόβλημα, θα ήθελα να σχολιάσω το έγγραφο αυτό. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 5, για την εισαγωγή ορίων στις απαιτήσει ε, που συζητήσαμε εδώ, θα πρέπει να παραμένουμε πιστοί στα κεφάλαια 4 και 5 θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί ενό γράφου που να αποτελεί και να προσφέρει προς τη θέμανια αξία στου καταναλωτέ. Και επίσης να είναι χρήσιμο και στη βιομηχανία. Το άρθρο 5 μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με κάποιες μικρές ελαφρές τροποποίησεις. Εάν συγκρίνουμε το κείμενο αυτό με την οδηγία περί υπηρεσιών, θα διαπιστώσουμε ότι το κείμενο εδώ είναι απλούστερο. Το άρθρο 5 λοιπόν μας επιτρέπει να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση που αυτή τη στιγμή μας λείπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και σε ένα κείμενο χρήσιμο και για τους καταναλωτές και για τη βιομηχανία. Τώρα για τις ε, οικονομικές υπηρεσίες, τις χρηματοπιστωτικές επίσης, εδώ νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο τομέα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα. Υπάρχει η δυνατότητα να επιφέρουμε μεγάλε αλλαγέ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τουλάχιστον ένα ελάχιστο όριο προστασία. Αυτό ήδη θα είναι μια επιτυχία. Σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη που έχουν ε, προβλέψει διατάξει για αυτό το τομέα, εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει αντίφαση νομική τουλάχιστον. Θα μπορούσαν να συνεχίζουν να εφαρμόζουν του δικού του κανόνε, του ειδικότερου κανόνε. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να στοχεύσουμε την ενιαία αγορά και μέτρα που να την ευνοούν. Νομίζω θα συνεννοηθούμε καλά και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την καλή συνεργασία. Ιδιαίτερα από την πλευρά του συντάκτη της έκθεσης. Ευχαριστώ. Uh, thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπίλαν. Ε, πρόεδρε, σε αυτό το στάδιο ασφαλώς δεν έχω μελετήσει τα δύο papers, αλλά βρίσκω αυτά τα οποία έχει πει ο Άντρεας πάρα πολύ λογικά και I could agree with them all the way. so we'll have more to say after we study the papers. Thank you. Uh, good. I think um, were there any other members who wanted to comment? Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι ε, συνάδελφοι που θα ήθελα να λάβουν το λόγο, ε, θα μπορούσα να πω εγώ την άποψή μου για το δεύτερο έγγραφο σχετικά με τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε σε ό,τι αφορά τι απαιτήσει ενημέρωση συγκεκριμένα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία τίθενται στο κείμενο. Βέβαια, για πρώτη φορά το βλέπουμε. Το, ε, το διάβασα όμω έτσι γρήγορα γρήγορα και είδα τα βασικά πορίσματα. Μιλάει για αλληλεπίδραση που δεν είναι βέλτιστη ιδίως ό,τι αφορά τις συμβάσεις, ε, κάνει λόγο για αλληλοεπικαλύψη αλλά και για κενά. Δεν ε, έχω καταλάβει ποια ακριβώς είναι η άποψη του εισηγητή για όλο το ζήτημα αυτό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να βγουν εκτό εντελώ οι υπηρεσίε αυτέ και άλλοι θεωρούν ότι απλά υπάρχουν κάποια κενά. Θα ήθελα να μα δώσετε κάποιε ενδείξει. Τι ε, αντίποση έχετε εσεί, αν έχετε διαβάσει αυτό το ενημερωτικό έγγραφο και εάν μπορείτε να μα κάνετε κάποιε συστάσει ήδη από τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας σταμάζω πραγματικά που παράλληλα και με άλλα πράγματα που κάνετε διαβάζετε και τη μελέτη. Ε, πρόκειται για το εξή, ε, για τις ε, τραπεζικές συναλλαγές. Για αυτές δεν υπάρχει επικάλυψη. Η δυσκολία έγκυται σε ασφαλιστικά συμβόλαια τα οποία συνάπτονται off-premises. Για αυτά δεν υπάρχει η ρύθμιση ανάκλησης. Δεν υπάρχει δίκαιο περί ανάκλησης αυτών των συμβολέων. Όμως τα ασφαλιστικά συμβόλαια παρουσιάζουν κάποιες ιδιομορφίες ε, που πρέπει να τις ε, λάβουμε υπόψη. Παραδείγματος χάρη, όσον αφορά στην ασφάλιση των αυτοκινήτων, ήδη την πρώτη μέρα πρέπει και αρχίζει να ισχύει το συμβόλαιο, ε, δεν είναι δυνατόν πλέον να ανακληθεί αυτή η υποχρέωση γιατί αρχίσει όπως σας είπα να τρέχει η κάλυψη, η ασφάλεια. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν, είναι, δεν λέω ότι δεν είναι σκόπιμο να επέμβουμε, όμως είναι υποχρέωση της Κομισιόν να ρυθμίσει, να ρυθμίσει αυτό το θέμα με ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση. Αν θέλετε μπορούμε και εμείς να συμπεριλάβουμε ε, ένα ε, εδάφιο Πάντως δεν θεωρώ ότι θα μπορέσουμε στο σημείο αυτό να επιτύχουμε ένα σαφή διαχωρισμό. Και γνωρίζω ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό και στη διαβουλεύση του Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν κρίνω ότι είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί επί του θέματος ο Μίχαλ Άντενχοφ. Ωραία. Νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να μελετήσουμε πιο εντελεχώς αυτά τα έγγραφα Όσοι δεν είναι εδώ σήμερα, πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να βρείτε αυτά τα έγγραφα στο, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, αλλά θα υπάρχουν ε, συνδέσεις και από την εσωτερική μας ιστοσελίδα, οπότε μπορείτε να μελετήσετε αυτά τα δύο έγγραφα από εκεί. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τι έχει να πει το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο υπήρξαν και κάποιε σημαντικέ εξελίξει ό,τι αφορά την άποψή του για το πώ θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η οδηγία. Ο κ. Βίλαν το ανέφερε, μίλησε νωρίτερα για το κεφάλαιο 5, μίλησε για την αξία προ καταναλωτέ κτλ. Ο κ. Έτενχοφ θα μπορούσε καταρχά να μα κάνει μια ενημέρωση και μετά ο κ. Πέτρου την Επιτροπή. Φαντάζομαι μετά θα ήθελε και ο εισηγητή να σχολιάσει και ίσω και οι συντάκτε τροπολογιών να χαιρετήσω τον κύριο Άτοχο και να τον παρακαλέσω να μας ενημερώσει για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και κυρίως και για το τι έγινε αυτό στην Κορεπέρ. Μπορώ να μιλήσω Ολλανδικά. Α, ωραία. Λοιπόν, όπως είπατε, πραγματικά συνέβησαν σημαντικά πράγματα στο Συμβούλιο. Χθε στην Κορεπέρ καταλήξαμε σε συμφωνία για την οδηγία αυτή, αλλά πρέπει να σας πω ότι πρέπει και να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Η συμφωνία προς το παρόν είναι στο επίπεδο της ε, Κορεπέρ. Παρακαλώ, πώς μπορείτε να αλλάξετε αίθουσα, παρακαλεί το ομιλητής, μάλλον ε, θέση. Ωραία, τώρα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να τα ξαναπώ από την αρχή. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Πράγματι λοιπόν συνέβησαν όπως είπατε και εσείς κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Φτάσαμε στην Κορεπέρ χθε σε συμφωνία η οποία όπως είπα πρέπει να εγκριθεί φυσικά και από το Σύμβουλο. Αυτό πρέπει να το καταστήσω σαφές. Ποιο είναι το αδρό περίγραμμα της συμφωνίας, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της συμφωνίας για την προσέγγιση σε σχέση με τα διάφορα κεφάλαια. Πρώτα απ' όλα επιλέξαμε να εστιάσουμε στις συμβάσεις ε, εξ αποστάσεως και ε, τα κεφάλαια 4 και 5 διαγράφηκαν από το Συμβούλιο. Δεδομένης της ελάχιστης εναρμόνισης η οποία υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία είτε για τους καταναλωτές είτε για την κυβέρνηση. Αποφασίσαμε λοιπόν να διαγράψουμε αυτά τα δύο κεφάλαια. Σε ό,τι αφορά τα δύο συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία συζητείτε σήμερα στην Επιτροπή σας, μπορώ να σας πω εμείς πώς ε, τα αντιμετωπίσαμε στο Συμβούλιο. Συγκεκριμένα εστιάσαμε σε αυτές τις δύο κατηγορίες ε, συμβάσεων και διατηρήσαμε τα κεφάλαια 1 και 3. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν θα συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής και σε ό,τι αφορά το κοινοτικό κεκτημένο, την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία δηλαδή, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν εδώ κάποιες δυσκολίες. Τομεακή κάθετη νομοθεσία, θέλουμε να προστατεύσουμε τα ε, δικαιώματα των ε, καταναλωτών που θεωρούνται λέξη γενεράλης. Και τώρα η οδηγία για τις υπηρεσίες και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο λαμβάνονται υπόψη ε, στον τομέα της. Η καθεμία βέβαια υπάρχουν κάποιες αλληλοεπικαλύψεις, αλλά θεωρεί το Συμβούλιο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και τις τρεις οδηγίες χωρίς να χρειαστεί τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 22.5 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, το οποίο καθορίζει ότι οι παρέχοντες υπηρεσίες, οι οποίοι είναι κατεστημένοι σε συγκεκριμένη επικράτα, μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες περιφέρειες. Δεν θα θέλαμε να υπάρχει καμία σύγκρουση ή αντίφαση στο ε, μέλλον. Η άποψη του Βελγίου είναι ότι προς το παρόν ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια ε, σύγκρουση διατάξεων, αλλά εάν αυτό συμβεί στο μέλλον θα υπάρξει σχετικός κανόνας, οπότε η οδηγία καταναλωτών θα υπερτερεί τον άλλον. Έτσι θεωρούμε ότι πρέπει να είναι σχέση μεταξύ των οδηγιών και με αυτόν τον τρόπο αποφασίσαμε να δώσουμε και τη ρυθμιστική μορφή σε αυτή τη διάταξη. Η τελική μορφή θα εγκριθεί από το Συμβούλιο, όπως σας είπα, αλλά σε ένα διαφορετικό σχηματισμό του Συμβουλίου και θα δημοσιευτεί και τότε. Thank uh, Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας παρουσιάσετε τις απόψεις του Συμβουλίου, διότι προφανώς είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Διότι και το Συμβούλιο περιμένει να δει πώς και η Επιτροπή θα κινηθεί σε αυτόν τον τομέα. Απλώς να μου διευκρινίσετε το εξή. Στο Συμβούλιο και επειδή βρισκόμαστε στην πρώτη ανάγνωση στη διαδικασία τη συναπόφαση. Οπότε θα πρέπει να έχετε και τη δική μα τοποθέτηση. Υποθέτω ότι βάσει όσων είπατε, η αρχική πρόταση τη Επιτροπή, που αρχικά θα καταργούσε την οδηγία για τους θέμετους όρους τους συμβασιακούς και την οδηγία για τις υπηρεσίες αυτές οι προτάσεις θα παραμένουν απαράλλατες. Οπότε η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών θα επικεντρώνεται πλέον στην αντικατάσταση των οδηγιών για τι πωλήσει από απόσταση και κατοίκων. Σωστά. Ωραία. Νομίζω ενδιαφέρον θα ήταν να ακούσουμε τι απόψει και τη επιτροπή, Διότι σε σχέση με την αρχική πρόταση τη Επιτροπή, εδώ οι αλλαγέ είναι αρκετά δραματικέ. Υπάρχει, θα έλεγα, δραματική απόκληση απόψεων μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπή. Δεν έχει αποφασίσει το κανεί ποια κατεύθυνση ακριβώ θα ακολουθήσει. Θα ήθελα όμω να ακούσω ποια είναι η αίσθηση και τη Επιτροπή για κάτι που θεωρώ ότι είναι μια αποφασιστική αλλαγή σε σχέση με την αρχική πρόταση τη Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν σημαντικά όσα είπε το Συμβούλιο. Θέλω να τα σχολιάσω πριν περάσω στα έγγραφα. Πρώτα απ' όλα, η Επιτροπή καλωσορίζει τη σκληρή και αποτελεσματική δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας. Δουλειά που μας επέτρεψε να πετύχουμε ιδιαίτερη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την Οδηγία περί καταναλωτών. Αυτό είναι πραγματικά άξιο να το σημειώσουμε. Έπειτα, Κάτι που επίσης αξίζει να τονίσουμε είναι ότι η Επιτροπή θα τοποθετηθεί οριστικά επί της συμβαστικής λύσης όταν προχωρήσουν και οι συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Και μάλιστα όταν περατωθούν στην πρώτη ανάγνωση. Δεν έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποια διαμορφωμένη άποψη σε σχέση με την ε, συμβιβαστική πρόταση του Συμβουλίου. Ωστόσο αναγνωρίζουμε το εξή. Το Συμβούλιο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα διέξοδο. Και η μόνη διέξοδος που εξήβρε ήταν να επικεντρωθεί σε μια σημεία της πρότασης στις διαπραγματεύσεις. Από αυτήν λοιπόν την άποψη, το κείμενο που συμφωνήθηκε στο επίπεδο του Κορεπέρ φαίνεται να αποτελεί μια βάση εργασίας ικανοποιητική προκειμένου να βελτιώσουμε με τα μέτρα που θα προβλέψουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λυπόταν εάν δεν πετυχαίναμε, μάλλον αν πετυχαίναμε συμφωνία με πλήρη εναρμόνιση των κεφαλαίων 4 και 5. Ωστόσο, το να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην πρόταση του Συμβουλίου ίσως είναι μια πρώτη οδός που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε και βέβαιοι πριν φανεί ποια είναι και εδώ η καλύτερη λύση. Στο τέλος της διαδικασίας θα δούμε τι τροπή θα έχουν πάρει οι συζητήσεις και πώς και εμείς θα τοποθετηθούμε. Σε ό,τι αφορά τα δύο ζητήματα που τέθηκαν εδώ, σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία, το ενημερωτικό σημείωμα για τη σχέση με την νομοθεσία νομίζω ε, συμμερίζεται το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε και στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ της οδηγίας δικαιωμάτων των καταναλωτών και της οριζόντιας νομοθεσίας, όπως της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη οδηγίας για τις υπηρεσίες, η σχέση αυτή θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νομοθέτημα θα πρέπει να ισχύει πλήρως εντός του ορισμένου πεδίου που προβλέπεται γι' αυτό. Δηλαδή και η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και για το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι δύο θα πρέπει να διέπονται από τις ίδιες υποχρεώσεις για ενημέρωση και οι δύο να εφαρμόζονται δύο κείμενα. Εφόσον υπάρξει σύγκρουση μεταξύ τους, διαφορά, η λογική λύση θα ήταν να υπερισχύσει οδηγία για τα δικαιώματα των καταλωτών. Αυτό ήταν το συμπέρασμα και του Συμβουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ το έργο του Συμβουλίου ως προς την νομοθεσία έδωσε λίγο πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θα είχαμε προτιμήσει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως πλήρη εναρμόνιση και σε τομείς όπου η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η οδηγία για, τα, για τις υπηρεσίες εφαρμόζονται. Δυστυχώς αυτό δεν το πετύχαμε. Δεν είχαμε αυτή τη συμφωνία στο Συμβούλιο. Κατά δεύτερον, για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και το σχετικό ζήτημα. Ο στόχο τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν να καλύψουμε τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε στο βαθμό κατά τον οποίο ούτω ή άλλω καλύπτονταν από την προϋπάρχουσα νομοθεσία το Ρίκας δηλαδή, που έγινε μέσω της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Προκειμένου να μην χάσουμε επίπεδα προστασίας που ήδη προβλέπονταν προηγουμένως. Γι' αυτόν τον λόγο, κυρίως για το κεφάλαιο 3, για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις συμβάσεις για τις εγκαταστάσεις, ε, εδώ ε, τα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ισχύουν μόνο για τι ε, εγκαταστάσει και για να διασφαλίσουμε την προστασία, ιδίω σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο για τις πιστώσει ε, των καταναλωτών. Δηλαδή συμβάσεις εκτών εγκαταστάσεων ή υπόθηκα δάνεια. Εδώ θα Είμαστε εκτός πεδίου. Επίσης ε, μιλάμε και για την ασφάλιση. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν να, μείνει εκτός η ασφάλιση, διότι εν μέρη καλύπτεται από τον μηχανισμό για την προστασία των καταναλωτών. Ιδίως ό,τι αφορά τις ασφάλειες ζωής, που κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσέφεραν επαρκή προστασία. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσει στο Συμβουλίο, όπω εξήγησε ο κ. Σέντεχοφ, οδήγησαν στην εξή κατάσταση. Δεν ήταν δυνατόν να παραμείνουμε στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εντός του πεδίου του κεφαλαίου 3. Η Επιτροπή λυπάται που δεν το πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank you both very much. I think... Ευχαριστώ και τους δυο σας. Νομίζω ότι ιδίω με βάση το Επιτροπή Συμβούλιο θέλω να παρακαλέσω τον εισηγητή. Α, θέλει να περιμέ... θέλετε να απαντήσετε, να περιμένουμε λίγο. Εντάξει, κύριο Λέχνερ, άλλοι ομιλητέ, άλλοι συνάδελφοι. Σε σχέση με την προσέγγιση του Συμβουλίου ή με τις δικές σας απόψεις, σε σχέση με τις δικές σας απόψεις. σε ό,τι αφορά τις σημαντικές αλλαγές στην πρόταση. Διαγραφή κεφαλαίου 4, κεφαλαίου 5, οι συμβάσει εκτός εγκαταστάσεων off-premises, ο Ανδρέας Φαπ, ο Κόρτ Λέχνερ, υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Άλλος ένας, ωραία. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον εισηγητή πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η Βελγική Προεδρία το δικό μου, τη δική μου την πρόταση ε, να συμπτυχθούν τα κεφάλαια 2 και 3 την υιοθέτησε. Και στο Συμβούλιο πέτυχε και την πλειοψηφία περί σύμπτυξη, για αυτή τη σύμπτυξη των κεφαλαίων 2 και 3. Αυτό λοιπόν πολύ σημαντικό και δείχνει ότι το Κοινοβούλιο σε αυτό το τόσο δύσκολο νομικό θέμα πέτυχε μια πολύ καλή συνεργασία. Όσον αφορά την διαγραφή των κεφαλαίων 4 και 5, σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να το πούμε αυτό εδώ γιατί η συνάδελφος κυρία Γκέπχατ και ο συνάδελφος Ροσφό δεν είναι σήμερα ο και Στούρνα και είπαμε ότι στο τέλος θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι στο Συμβούλιο όσον αφορά το άρθρο 22 και τη μετακύληση του κινδύνου που εμπεριέχει το άρθρο 23, επ' αυτόν επιτεύχθηκε συμφωνία. Έτσι λοιπόν τίθεται το εξή ερώτημα, κατά πόσον η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί και σε όλες τις συναλλαγές και ενδεχομένως τα πράγματα να γίνουν διαφορετικά από αυτά που λέει το ε, Συμβούλιο, δηλαδή να ισχύουν μόνο για τα κεφάλαια 2 και 3. Και στην περίπτωση αυτή θα είχαμε διαφοροποίηση των προϋποθέσεων παράδοσης και των προϋποθέσεων μετακύλης του κινδύνου σε συμβόλαια εκτός εγκαταστάσεων off-premises. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Θα μπορούσε λοιπόν να προκύψει πρόβλημα. Θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε και σε επίπεδο σκιωθών εισηγητών στην Επιτροπή μας και μετά θα αποφασίσουμε. Γενικά θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι η Βελγική Προεδρία ε, θεωρεί ότι το Συμβούλιο μπορεί να συμφωνήσει με αυτού του θέματος και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα και για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ε, την τελευταία φορά τοποθετήθηκα. Ε, την προσέγγιση του Συμβουλίου την βρίσκω απόλυτα λογική. Ε, δεν νομίζω ότι αλλιώς μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η οδηγία. Το είπα και την τελευταία φορά. Οι δικέ μου ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω κάτι για την σημερινή πρόταση. Κοιτάξτε, το ε, πώς ακριβώς ε, συσχετίζονται οι οδηγίες ή τα νομοθετικά κείμενα, νομίζω είναι αυτονόητο ότι όταν κατατίθεται μία οδηγία θα πρέπει να υπάρχει αυτή η αρμονία. Δύσκολο βέβαια, αλλά ε, καταρχήν πρέπει κανείς να δει τι λέει το επόμενο κείμενο, ποια είναι η βάση πάνω στην οποία εργαζόμαστε. Αυτό είναι αυτονόητο και δεν είναι καθήκον του Κοινοβουλίου να το πράξει αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω και αναφέρομαι εδώ στα θέματα ουσίας περί των οποίων πρόκειται. Ε, μέχρι τώρα δεν υπήρξε ούτε αιτιολόγηση ούτε εξήγηση. Ο συνάδελφος κ. Σβάπ μίλησε για την παράδοση των εμπορευμάτων. Πότε προκύπτει κίνδυνος στην αγορά ο κίνδυνος εμφανίζεται κατά την αγορά ή κατά την παράδοση. Αυτό είναι καθοριστική σημασία σε ένα συμβόλαιο και δεν υπάρχει καμία αιτιολογία. Δηλαδή εκπονείται ένας κανονισμός χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια έρευνα. Είναι σωστός ο κανονισμός. Τι γίνεται στις διάφορες χώρες. Ε, τι είδου συνέπειες θα προκύψουν. Ο κύριος Σβάπ το ανέφερε αυτό και ε, το να προκύπτει σε ένα τέτοιο ερώτημα το ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει έρευνα, αυτό είναι αυτονόητο. Η Κομισιόν δεν το έπραξε, το παρέλειψε. Τουλάχιστον για αυτά τα ερωτήματα και υπάρχουν τουλάχιστον 30 τέτοιου είδου ερωτήματα στο κείμενο, να υπάρχει λοιπόν αιτιολογία, έρευνα, συζήτηση. Κατά την άποψή μου δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άλλο δρόμο. Εκτός και αν διαφωνεί ο εισηγητής, ο κύριος Λέχνερ, νομίζω θα παραδεχτεί ότι υπάρχει ένα πολύ διεξοδικό διάγραμμα. Σε εσά απαντώ. Όπως θύμισα εδώ, έχουμε μια διεξοδική ανάλυση που μας ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, διαφορές και ιδίως για τον ε, κίνδυνο που προκύπτει σε κάθε διαφορετική χώρα. Αυτά ήδη υπάρχουν. Τόσο λοιπόν εδώ και με διαψεύσιο ο εισηγητής. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε ε, Περισσότερε πληροφορίε για αυτά τα ζητήματα. αποφάσει πρέπει να λάβουμε. Ο κύριο Μάντερ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Λυπούμε που έχει αποδυναμωθεί η πρόταση με τη διαγραφή των κεφαλών 4 και 5. Αν όμω αυτό είναι ο μόνο τρόπο επίτευξη συμφωνία, σα βελτιωθεί ένα μικρό τμήμα τη πρόταση από το τίποτα. Σε ό,τι αφορά τη χρονομίστωση, επειδή ήμουν εισηγητή, ε, γνωρίζω ότι υλοποιείται σε διάφορα ε, επίπεδα. Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει σε ποια χώρα αγοράζει ή μπορεί να το γνωρίσει αλλά δεν, γνωρίζουμε πώς εφαρμόζεται, δεν γνωρίζει μάλλον πώς εφαρμόζεται η οδηγία. Λοιπόν, διαγραφούν τα κεφάλαια 4 και 5. Νομίζω ότι καλό θα ήταν, ε, μπορεί ο Αντρέας να το συμπεριλάβει αυτό. Μήπως η οδηγία πρέπει να γίνει κανονισμός ώστε πραγματικά να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών. Αυτό άλλωστε συμβουλεύει και ο Μόντι. Ελπίζω όλοι αυτοί να ακούν και ίσως να εκμεταλλευτούν τα Χριστούγεννα όπως και εμείς για να το σκεφτούμε καλύτερα το όλο θέμα. Γιατί αν θέλουμε να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά αυτό θα πρέπει να δούμε και να μην μιλάμε για τα εθνικά συμφέροντα. Okay, well, I'm going to close the discussion now, Εδώ θα λήξει η συζήτηση. Εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς. Άρα με το νέο έτος θα τα ξαναπούμε για το θέμα αυτό. Είμαστε στην πρώτη ανάγνωση. Είναι πολύ κρίσιμη λοιπόν η θέση του Κοινοβουλίου. Μας ενδιαφέρουν και οι απόψεις βέβαια του Συμβουλίου. Ο κύριος Βάπ φαντάζομαι ότι θα μας προτείνει και τις ιδέες του για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μέχρι την ψηφοφορία του Ιανουαρίου. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στην έναρξη μιας διαδικασίας, στον αρκτήριο λάκτισμα, θέλετε, μιας πολύ σημαντικής ε, ε, πράξης που προτείνεται για την ενιαία αγορά. Ξέρετε ότι έχουμε αποφασίσει να εξετάσουμε αναλυτικά με την ε, εκπόνηση τριών εκθέσεων την προτινόμενη πράξη για την ενιαία αγορά. Προτάσεις για καθένα από τα τρία κεφάλαια της πράξης για την ενιαία αγορά. Έχουμε λοιπόν τα τρία κεφάλαια. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά. Ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους. Ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Αυτά είναι τα τρία κεφάλαια. Δύο από τους τρεις εισηγητές είναι παρότες. Κυρία Κανιέτη ασχολείται με τη διακυβέρνηση. Ο καθηγητής Κορέα Κάμπος ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους. Αλλά ο κύριος Μπουζόη επειδή θα υποστηρίξει το δακτορικό του σήμερα, θα είναι δόκτωρ όταν επανέλθουμε μετά τις γιορτές, θα μας πει ο κύριος Μπουζόη τότε τι πιστεύει, θα τον αντικαταστήσει όμως ένας άλλος συνάδελφος. Έχουμε κάποιο χρόνο για τη συζήτηση, δεν είναι όλοι συγητές. Θα ρωτήσω το εξής τους συγητές. Εγώ σας παρακαλώ να παρουσιάσετε ο ένας μετά τον άλλο, οι δύο που είστε εδώ, και ο τρίτος παντικαθιστά ε, τις ε, προτάσεις, τα σκέλη ο καθένας που έχει αναλάβει για να έχουμε μια γενική εικόνα για την προτινόμενη αυτή πράξη και στη συνέχεια θα ζητήσω από τους σκιώδεις εισηγητές να μιλήσουν και αυτοί. Δεν χρειάζεται να πάμε με τη σειρά, τις τρεις εκθέσεις, μπορεί κάποιος σκιώδης να μιλήσει για τη μία, για την άλλη, δεν έχει σημασία η σειρά. Κανιέτη, Κορέα Κάμπος, Κρόιτσμαν είναι τρει πρώτοι οι συγητέ μας. Η κυρία Κανιέτη νομίζω έχει και κάποια slides, κάποιες διαφάνεις να μας παρουσιάσει. Λοιπόν, σα δίνω το λόγο και ξεκινά λοιπόν εδώ η συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ η διακυβέρνηση τη ενή αγορά μα ενδιαφέρει από την άποψη του πώ θα διαθέσουμε υπηρεσίε στους πολίτε και πώ θα τη διακυβερνήσουμε αυτή την αγορά προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και να ωφεληθούν οι πολίτε. Δεν βλέπω τίποτα στην ε, οθόνη. Λοιπόν, πρώτη διαφάνεια, στόχοι. Ένα από τα ζητήματα που το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει και να καθορίσει είναι ποιε είναι οι φιλοδοξίε μα για την πράξη της ενιαίας αγοράς. Θα ενισχύσουμε την ενιαία αγορά, θα προσθέσουμε, θα κάνουμε και άλλα βήματα προς τη διαδικασία της ενοποίησης. Αυτό ζητώ εγώ να μάθω εδώ στην πρώτη διαφάνεια. Πρώτα απ' όλα να ορίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, διότι μεταξύ των διαφόρων προτάσεων των 50 περίπου θα πρέπει να διαλέξουμε 12, 15 ως τις πρώτες που θα θέλαμε να υλοποιηθούν ως μέτρα. Έπειτα πρέπει να καταδείξουμε και την προτιμόμενη κατεύθυνση καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα για τις ε, πρωτοβουλίες προτεραιότητας που θα πρέπει να αναλυθούν ως το 2012. Έπειτα το θέμα είναι αν θα προτείνουμε και επιπλέον πρωτοβουλίες στην ε, πράξη της ενιαίας αγοράς και αν μπορούμε να προτείνουμε και βελτιώσεις. Επίσης, αυτό που θεωρώ άκρο σημαντικό είναι να Βάσει των τριών πυλώνων της ενίας αγοράς, της διακυβέρνησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, βάσει αυτών των πυλώνων να καταρτήσουμε και την έκθεση. Και πρέπει να ακολουθήσουμε εδώ μια συνολική σφαιρική προσέγγιση. Μιλάμε για ένα πακέτο ε, ενιαίο, για μια ενιαία πράξη. Η νομοθεσία αφορά και τους τρεις πυλώνες και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Αυτά που βλέπω εγώ ως καθοριστικά ζητήματα τώρα. Σημεία κλειδιά Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το ρόλο της Επιτροπής ε, για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, για τη σύμπηξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων και των κρατών μελών. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε τι κίνητρα μπορούν να δοθούν για να υπάρχει έγκαιρη και σωστή εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Νομίζω ότι ε, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και βέβαια εν συνεχεία θα πρέπει να σκεφτούμε ποια ακριβώς είναι αυτή η πολυμερής προσέγγιση. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, πίνακες συσχέτησης, ε, πίνακες επιδόσεων, σκόρμπορς κτλ. Σε ό,τι αφορά δε την διαδικασία της αμοιβαίας αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνεται στην οδηγία της υπηρεσία, πώς μπορεί να εφαρμοστεί και θα πρέπει να δούμε επίσης πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και τη διοικητική συνεργασία στο πλαίσιο του συστήματος ε, ενδοκινοτικής ενημέρωσης ε, Solvit. Να περάσουμε παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ανταγωνιστικότητα της ε, Ένωσης είναι η βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τι εναλλακτικέ μορφέ επίλυσης διαφορών, κάτι που υπάρχει ήδη. Το solve για παράδειγμα, υπάρχουν 1.500 ε, υποθέσεις. Όμως οι πολίτε της Ένωσης είναι 500 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε στην αρχή. Εάν μιλήσουμε επίσης για τον χρόνο που παίρνει η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Πρέπει να δούμε πώς τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερο γιατί έχουν ένα ρόλο να διδραματίσουν και αυτά ε, στην ε, μείωση της, ε, του χρόνου που απαιτείται για τη μεταφορά του στο εθνικό δίκαιο. Ήδη εξετάζονται οι βέλτιστες πρακτικές ανταλλαγή βάση των πρακτικών. Πρέπει όμως ήδη, πρέπει να γίνουν περισσότερα, πρέπει να παροτρύνουμε να γίνουν περισσότερα. Και θα πρέπει και στην έκθεση να φαίνεται η παρότρινση αυτή. σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις, ό,τι αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, έχουμε κάποια ορόσημα, έχουμε κάποια benchmarks, σημεία αναφοράς. Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο χρόνος για τη συμμόρφωση προς αυτά τα σημεία. Διαβάζοντας την έκθεση, πραγματικά ξεπλάγει, βλέποντας πόσες μοναπευθυντικές θηρίδες υπάρχουν μία δίνει ενημέρωση, ε, άλλες βοηθούν τη διοίκηση να αντιμετωπίσει ιδέως συνοριακά ζητήματα. Θα πρέπει να μπορέσουμε κάπως να ενοποιήσουμε ε, αυτά τα one-stop shops, τις πολυάριθμες αυτές ε, μοναπευθυντικές θηρίδες. Τώρα, έκθεση Μόντι. Προτείνει ότι ένας πιθανός από τους τρόπους να εδρεωθεί καλύτερα η μια αγορά είναι πρώτα να σκεφτόμαστε για κανονισμούς και μετά για οδηγίες. Οι κανονισμοί βέβαια δεν θα επιλύσουν όλα τα προβλήματα, ωστόσο αυτή είναι η διέξοδος. Επίσης, ό,τι αφορά τους πίνακες συσχέτισης για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό ότι πολλά κράτη-μέλη ε, είναι ιδιαίτερα έχουν δισταγμού στο να παράσχουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τους πίνακες συσχέτιση και ίσω θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε να καταστήσουμε υποχρεωτική την υποβολή των στοιχείων για τους πίνακες συσχέτισης. Μία από τις ιδέες που θα πρέπει να εξετάσουμε μεταξύ μας εδώ είναι πώς θα μπορούσαμε να παράσχουμε ευρύτερη χρήση του, σχήμα, του σχήματος του 28 scheme, regime, που πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει. Το 28ο καθεστώ σύστημα. Επίσης, θα πρέπει να διατηρηθεί ολιστική και κοινή προσέγγιση στην ενιαία αγορά. παρότι έχουμε γνωρίζουμε τρεις εκθέσεις διαφορετικές. Θα γράψουμε λοιπόν τρεις εκθέσεις που σίγουρα θα βασίζονται σε προηγούμενες εκθέσεις Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. οι οποίες αναλύουν την ενιαία αγορά από συγκεκριμένα οπτικές γωνίες. Εγώ προσβλέπω στη συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές μια ομάδα στην οποία θα λάβουν μέρος και άλλοι συγητές. Και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω λίγο το χρονοδιάγραμμα. Η υποβολή των σχεδίων έκθεση από πλευρά μας 12 Ιανουαρίου. Εν συνεχεία εξέταση σχεδίων έκθεσης για το Φεβρουάριο, 1η Φεβρουάριο συγκεκριμένα, κατάθεση τροπολογιών 7 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 28 Φεβρουαρίου και ελπίζουμε στις 23 Μαρτίου στην Ολομέλεια να μπορέσουν να γίνουν δεκτές και οι τρεις εκθέσεις. Αυτό βέβαια θα απαιτήσει εξαιρετική πειθαρχία, αποφασιστικότητα, επιμονή, γιατί για τη διακυβέρνηση υπάρχουν 10 ακόμη επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένα τιτάνιο έργο μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και τη συζήτηση στις τέσσερις από τους μήνες μεταξύ των Ευρωπαίων και στο τέλος θα πρέπει όλα αυτά να τα συμπεριλάβουμε στην νομοθεσία που θα προκύψει ως απόρρια του δικού μας έργου. Ευχαριστώ. Well, Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ε, κάνατε μια τόσο καλή έναρξη ε, και ήταν και μια πολύ καλή ευκαιρία για να μας υπενθυμίσετε την ολιστική φύση αυτής της συζήτησης, πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, βεβαίως και έχετε δίκιο, έχουμε ένα ε, φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να συμπέσουμε με το τέλος της περίοδου διαβουλεύσεων και κυρίως εν τέλη Μαρτίου θα συνέλθουν οι Υπουργοί για να εγκρίνουν αυτή την πράξη. Συζήτησα βέβαια με τους προέδρους των επιτροπών που γνωμοδοτούν για το χρονοδιάγραμμα και καταλήξαμε στο ότι μετά τις 28 θα πρέπει να έχουμε με ειδική ημερομηνία για ψηφοφορία εφόσον βέβαια οι επιτροπές γνωμοδοτήσουν έγκαιρα. Εσείς ως εισηγητές θα έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε ε, τις ε, γνωμοδοτήσεις σας και ορισμένες επιτροπές συμφώνησαν ότι ε, είναι δική τους ευθύνη να καταρτήσουν κάποιες ε, προτάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας στείλουν οπωσδήποτε τα σχόλιά τους για να συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο. Ας περάσουμε τώρα στον ε, επόμενο μιλητή, στον καθηγητή Φερνάντο Ντε Κάμπος, θα πρέπει βέβαια να έχουμε μεταξύ και έναν κατάλογο μιλητών. Δεν ξέρω αν θέλουν να μιλήσουν ε, όλοι οι σκιώδει, ε, ίσω και κάποιο άλλο που δεν είναι σκιώδη ηγητή. Μπορούμε να βάλουμε τώρα το όνομά του στο κατάλογο για να το γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα εξή ονόματα μετά τον εισηγητή. Μετά τον εισηγητή έχουμε. Mrs. McClarkin, Mrs. Mrs. Um, I'm also a shadow, so I will have, have a, and, Mrs. Mrs. Και εγώ θέλω να μιλήσω, δεν ξέρω. Α, και η κυρία Τάιλερ. Σας ε, βάζω πριν από την κυρία Τούρναμ. Και η κυρία Τάιλερ λοιπόν, άλλοι συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλο να μιλήσει. Αν επιθυμεί μπορεί όμως να λάβει το λόγο. Καθηγητής ε, Ντεκάμπος, ε, μπορείτε αν θέλετε να μας μιλήσετε για την δεύτερη έκθεση, την ενιαία αγορά για τους ε, Ευρωπαίους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή είναι άκρο σημαντική για όλους μας, ιδίως για τους Ευρωπαίους. Έχει σχέση με δύο εκθέσεις, την έκθεση Γκρέκ και Μόντι, που μπορεί να θεωρηθούν ε, συγγενικές. Όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ θα πρέπει να επικεντρωθώ εγώ στο κεφάλαιο 2 της ανακοίνωσης για την, πράξη, για την πράξη της ενιαίας αγοράς με 21 προτάσεις. Αυτά θα πρέπει να σχολιάσω στην εκθέσή μου. Η προσέγγιση που θα ακολουθήσω ως εισηγητής αφορά δύο επιλογές κυρίως. Πρώτα απ' όλα το μέρος της αναγνώρισης του πόσο έχει οδηγηθεί σε κόπωση η ενιαία αγορά βάσει της έκφρασης Μόντι και επειδή οι προσπάθειες αυτές πρέπει να αφορούν περισσότερο την ε, αγορά και τη διοργάνωσή του παρά ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών και μόνο. Για να ακολουθήσουμε αυτή τη θεώρηση πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουν γίνει λίγες μελέτες αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη βασική κατεύθυνση είναι ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν είναι κάτι που οικοδομείται αυτορμήτως. Υπάρχει έλλειμμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Όμω η εμπιστοσύνη των πολιτών ακριβώ δεν είναι κάτι που δημιουργείται αυτομάτω. Πρέπει να γεννάται η εμπιστοσύνη, να χτίζεται, να ε, υποδαβλίζεται. Και επειδή ακριβώ δεν είναι αυτόματη, είναι μια συμφωνία άρρητη ε, μεταξύ των καταναλωτών. Άρα αυτό έχει και πρακτικές συνέπειες, χειροπιαστές. Έτσι μπορεί να γίνει η αγορά ενιαία και να συμμετέχουν οι πολίτες ακόμα και πιο ευαλώτοι, πιο ευαίσθητοι. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η οριζόντια κοινωνική ρήτρα που προβλέπεται και από την συνθήκη για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ο μόνος τρόπος να είναι εύρυθμη η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αφορά και την οικονομία και το πώς ε, ε, οι πολίτες συμμετέχουν στην αγορά. Θα πρέπει πάντοτε ο πολίτης να βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος. Δεν μπορεί να υπάρξουν καλές λύσεις στην εσωτερική αγορά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις για την απασχόληση, την ε, οικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον ή την εμπιστοσύνη των πολιτών που καταναλώνουν ασφαλή προϊόντα. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι οι δυσκολίες συμπερίληψης ε, οργάνων και νομοθετικών προτάσεων ή μηχανισμών. Είδαμε ήδη με την οδηγία που μόλις συζητήσαμε ποιες είναι οι διάφορες περιοχές που μπορεί να υπάρξει επικάλυψη. Εδώ δύο επίτροποι τουλάχιστον πρέπει να συνδυαστούν για να δώσουν ένα κοινό ρεύμα δράσης. Ε, εδώ θα πρέπει να είμαστε λοιπόν ε, φιλόδοξοι αλλά με υγιείς φιλοδοξίες και να διατηρούμε διαρκή τη μέρημνα για την επικέντρωσή μας στο συμφέρον των πολιτών. Εάν ο πολίτης δεν καταλάβει τις, ε, τα ωφέλη από τη λειτουργία της, της ενιαίας αγοράς θα την υποτιμήσει. Θα υποβαθμιστεί η προσπάθεια. Έχουμε πολύ καλά παραδείγματα από το παρελθόν για το φαινόμενο αυτό. Τώρα, πώς θα προσπαθήσουμε να υπερβούμε το πρόβλημα της έκφρασης των προτάσεων και της αλλαγής προτεραιοτήτων. Στο κεφάλαιο 2 και σε σχέση με τις προτάσεις που γίνονται εκεί, ε, έχουμε άμεσες συνέπειες για τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια μελέτης, δημιουργώντας ένα πίνακα αποτίμησης με πέντε μεταβλητές. Η, η πρώτη είναι η προτινόμενη μορφή παρέμβασης, δηλαδή ένα νομοθέτημα ή μια δράση ή μια απλή ενημέρωση. Η μορφή παρέμβασης θα πρέπει ακριβώς να μας δώσει μια κατεύθυνση για το μελλοντικό μας έργο. Η δεύτερη μεταβλητή είναι το πόσο χειροπιαστά θα είναι τα αποτελέσματα για τους πολίτες. Είναι χρήσιμα, είναι χειροπιαστά τα αποτελέσματα των μέτρων που προβλέπονται. Πρέπει να μπορεί ο πολίτη να τα αγγίξει για να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνη. Η τρίτη μεταβλητή είναι η, πλήρωση της, η, κάλυψη μάλλον τη οριζόντια κοινωνική ρήτρα. Η τέταρτη είναι να σκεφτούμε είναι η ημερομηνία θέση σε ισχύ. Ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά στο πρώτο εξάμεινο το 2012 ή αργότερα, αλλά θα παίξει ρόλο. Και μετά η πέμπτη μεταβλητή είναι το πόσο εύκολα θα περάσουμε στην πράξη. Αυτό το σχήμα με τι πέντε μεταβλητέ θα μα επιτρέψει να εντοπίσουμε ενδεχόμενα κενά ή ευάλωτα σημεία στι προτάσει μα. Πέραν τη υπολογιζόμενη αξία τη πρόταση. Τώρα θα θέλαμε να προτείνουμε στου κοιόδη συζητητέ μια μορφή συνεργασία για να επεξεργαστούμε μαζί αυτόν τον πίνακα μεταβλητών, ώστε να καταλήξουμε σε μεθόδου αναζήτηση ε, συνένεση, ε, για να αναζητήσουμε και τους στόχους των μέτρων αυτών. Με, τα, με τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε τρεις βασικούς τομείς. Να είναι χειροπιαστά τα αποτελέσματα των μέτρων, το χρονοδιάγραμμα και το πόσο ε, εύκολα θα είναι στην υλοποίηση τα μέτρα. Υπάρχουν μέτρα λοιπόν τα οποία δεν ε, είναι εύκολα να συζητηθούν αλλά είναι πολύ χειροπιαστά τα αποτελέσματά τους και το αντίστροφο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να αναζητήσουμε τα κατάλληλα μέσα παρέμβαση. Θα είναι νομοθέτημα αυτό που θα προβλέψουμε, μια απλή ενημέρωση. Οι διαφορές αυτές είναι σημαντικές και είναι κάτι που θα πρέπει να το διερευνήσουμε στη συζήτησή μας. Ως ε, προς το χρονοδιάγραμμα θα συμφωνήσω με την κυρία Καλνιέτα. Είναι πιεστικό αρκετά, αλλά θα πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί στην εργασία μας και πολύ φιλόδοξοι. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για το πολύ επικοδομητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ενταχθήκατε και ίσω θα επανέλθω και εγώ αργότερα με την ιδιότητά μου του σκιώδου εισηγητού. Κύριε Κρόιτσμαν, ε, τώρα θα μιλήσετε εξ ονόμου του κυρίου Μπουζόη ε, και θα ξεκινήσουμε μετά τη συζήτηση με τους σκιώδους εισηγητές. Ο κύριος ε, Κρόιτσμαν. Ο κύριος Μπουσόη πρώτα απ' όλα θέλει να ζητήσει συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα εδώ το είπατε κι εσείς. Ε, η έκθεσή του εντάσσεται μέσα σε ένα πακέτο με πολύ αυστηρόχρονο διάγραμμα. Θέλει λοιπόν να ανταλλάξει μαζί σας απόψεις για τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν έτσι ώστε οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη να μπορούν να υποφελθούν πλήρως από την ενιαία αγορά. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική σε αυτή την δύσκολη περιοχή που ζούμε και αν θέλουμε ανάπτυξη πρέπει να έχουμε μια ενιαία αγορά φιλική ε, προς τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι και το νόημα της ε, έκθεσης. Αναφέρεται λοιπόν το θέμα των, ε, της παροχής υπηρεσιών. Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη. Ο εισηγητής ε, αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων. Είναι ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Επιπρόσθετα μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός ε, στις επιχειρήσεις, στο ε, εμπόριο ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται οπωσδήποτε την ενιαία αγορά. Και αυτό για να μπορέσει η Ευρώπη να συναλλάσσεται με άλλες ε, χώρες ε, του κόσμου. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μικρότερη ανάπτυξη από τις ΗΠΑ, αυτό οφείλεται εν μέρη και στο ότι δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ενέχει τεράστιες δυνατότητες. Η Κομισιόν λοιπόν πρέπει να διευκρινίσει το πλαίσιο που καθορίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο και εφόσον υπάρχουν δυσκολίες σε εθνικές ρυθμίσει που παρεμποδίζουν το εμπόριο αυτό, να τις εξελίψει. Πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη στο εμπόριο αυτό, όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις ε, που κάποιες φορές ε, είναι διστακτικέ στο να καταφύγουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να διευκολύνουμε και την ε, ανάκτηση χρέους γιατί αυτό πολλές φορές παρεμποδίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τελικά ε, εάν αναπτυχθεί αυτό το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μειωθεί το διοικητικό κόστος ε, κυρίως όταν είμαστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό η συγητής πιστεύει ότι υπάρχει μια πρόταση της αμοιβαίας αναγνώρισης ε, περί ταύτισης και εξακρίβωσης της γνησιότητας. Υπάρχει και μια ρυθμίση σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή. Αυτά τα στοιχεία είναι καθοριστική σημασία μια άλλη προτεραιότητα που αναφέρεται στην έκθεση είναι το να στηριχθούν οι επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους για καινοτομίε. Η νέα αγορά πρέπει να στηρίζει όλες τις επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδοθεί σε αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την καινοτομία και δεν μπορούν να υποφεληθούν πλήρω από την ενιαία αγορά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι κινητήρια δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρουν πολλές θέσεις απασχόλησης, αλλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και αυτό τους δημιουργεί δυσκολίες. Ο δυναμισμός επίσης επηρεάζεται ερνητικά από το διοικητικό φορτίο το οποίο πρέπει να περιοριστεί. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να χρηματοδοτηθούν μέσα από την κεφαλαϊκή αγορά και η Κομισιόν ε, είναι πρόθυμη να το υπογραμμίσει αυτό. Η Κομισιόν λέει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η παρουσία των εισηγητών, των να για τους επενδυτές οι ε, μικρομεσαίες πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα τις ε, ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά, όπως επίσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία ε, Επιπλέον, ε, θα πρέπει να διευκολυθούν περαιτέρω οι καινοτομίε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να βελτιώσει την ε, δυνατότητα συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ερευνητικά προγράμματα. Υποστήριξη λοιπόν της καινοτομία όχι μόνο για τις μικρομεσαίες αλλά για όλες τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό ο εισηγητής ε, συμφωνεί με τα ομολογιακά δάνεια να εκδοθούν αυτά από την ιδιωτική αγορά γιατί έτσι θα καταστεί να συγκεντρωθούν πόροι. Η Κομισιόν ε, πρέπει να καταστήσει σαφές ε, ότι οι διαδικασίες ε, για αυτά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι κατάλληλες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τέλος, ο εισηγητής χαιρετεί την πρόταση Κομισιόν να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στο venture capital να επενδύσει σε όλα τα κράτη-μέλη. Το venture capital, το επιχειρηματικό αυτό κεφάλαιο, κεφάλαιο είναι χρήσιμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να επικεντρωθεί σε καινοτόμου τομεί εάν η ενιαία αγορά δεν θα προσφέρεται και για το επιχειρηματικό κεφάλαιο, το venture capital ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές χρειάζονται και μια νέα αγορά για τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Πρέπει να διευκολύνεται η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαδικασία περί δημοσίων συμβάσεων. Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ε, σημασία στην ε, εξωτερική διάσταση των δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή η δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ξένες αγορές. Αν θέλει κανείς να είναι ανταγωνιστικός, δεν πρέπει να ε, περιορίζεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει να ε, δίδει μεγαλύτερη σημασία στις εξωτερικές συναλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη μόχλευση για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Τα φορολογικά μέτρα είναι πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό, πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ προσεκτικά. Ο συντονισμό των φορολογικών πολιτικών και εισαγωγή ενό ε, ενιαίου ε, εταιρικού φόρου δεν είναι κακή ιδέα. Το πλεονέκτημα βέβαια θα ήταν ότι οι επιχειρήσει Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια και θα είναι εύκολο να συγκρίνει κανεί ε, για τους διάφορες, τα διάφορα φορολογικά μέτρα που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Από την άλλη πλευρά αυτό δεν είναι το μόνο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν ε, να ε, έχουν ε, διαστηνοριακές συναλλαγές. Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο ο εισηγητής ήθελε να έχει την άποψη και άλλων πολιτικών ομάδων. Από την άλλη στηρίζει την ε, δημιουργία μιας νέας στρατηγικής ΦΠΑ που θα επιτρέπει να προσαρμοστεί το πλαίσιο στη νέα πραγματικότητα των οικονομιών πραγματικότητα που θα αποφέρει όφελο στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι κανονισμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη του. το ειδικό βάρο που υπάρχει για τι επιχειρήσει, τα εμπόδια που υπάρχουν στις διασυνοριακές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτέ λοιπόν είναι οι προτεραιότητε που έχει αντιμετωπίσει ο Κρίστιαν Μπουσόη. Είναι ανοιχτό βέβαια για συζήτηση και με μεγάλη του χαρά θα ακούει και τη δική σα την παρέμβαση για τα θέματα αυτά, αλλά ίσω και για άλλα που θέλετε μπορείτε να προβάλλετε. Η συνάντηση των συγητών, των σκιωδών, ε, σκιωδών με συγχωρείτε, θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Εκεί θα είναι δυνατόν να έχουμε μια ε, απευθεία ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εκπροσωπήσετε τον κύριο Μπουζόη. Ήταν ε, πολύ ξεκάθαρη δήλωση την οποία μας αναγνώσατε. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα για ανταλλαγή απόψεων, άρα δεν θα περιορίσω κανέναν να σας πω ποιοι είναι οι ομιλητές. We'll start with Mrs. Toon, Toon. Ripo, um, then... Um, Ripo. Μετά, δεν ξέρω, Τούρινεν Ρούλε, ποιος θέλει να ξεκινήσει, ποια θέλει να ξεκινήσει. Τούρινεν. Μακλάρκιν, Τρεταφυλίδης. Mrs. Ρούλε, um, Mrs. Styler, and I will also um, comment in my... Και θα μιλήσω και εγώ. γιατί με σκιώθησε για την ε, ενιαία χώρα για τους Ευρωπαίους και πρόεδρος βέβαια. Λοιπόν, κυρία τουρνέ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μάλκομ. Το πρώτο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι ότι χαιρόμαστε που υπάρχει και αυτό το έγγραφο για την ε, ενιαία πράξη, μάλλον για την πράξη για την ενιαία αγορά και βέβαια και όλες αυτές τις ε, εκθέσεις. Και συμφωνώ με την κυρία Καλνιέτα που είπε ότι είναι πολύ σημαντική ολιστική προσέγγιση. Όλοι πρέπει να εργαστούμε από κοινού. Έχουμε τρεις μεν διαφορετικές εκθέσεις, ένα όμως είναι το έγγραφο, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μία στρατηγική, ένα έγγραφο, άρα μεγάλη σημασία έχει η συνεργασία μας. Κάποιοι είπατε ότι υπάρχει κάποια κόπωση στην ενία αγορά. Ούτε το καταλαβαίνω, ε, ούτε το βλέπω. Γιατί εγώ έχω αντίθετα την εντύπωση ότι η ενία αγορά δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμη να λειτουργεί. Και αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει δεν είναι η κόπωση, είναι η αρχή. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν τώρα με την πολύ δυναμική προσέγγιση του τρόπου Μπαρνιέ δίνει ο κύριος Μπαρνιέ όθηση στην ενιαία αγορά. Είναι μια στιγμή που πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να προωθήσουμε τις εξελίξεις ε, στην ενιαία αγορά. Άρα εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη κόποση για την ενιαία αγορά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, θα είμαι σκιώδης για το δεύτερο σκέλος της πράξης για την ενιαία αγορά. Αν η ενιαία αγορά δεν αναπτυχθεί όσο γρήγορα θα θέλαμε και ελπίζουμε αυτό να συμβεί τώρα, εάν εγκρίνουμε τα σχέδια του Επιτρόπου Μπαρνιέ. Αυτό που θα χρειαστεί θα είναι η συμμετοχή όλων των πολιτών και όλων των ε, φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενιαία αγοράς. Όταν μιλάω για τους πολίτες, το έχω ξαναπεί στην Επιτροπή μας, ε, ουσιαστικά μιλώ για την ενημέρωση, έλλειψη ενημέρωση. Και αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πράξη ενιαία αγορά. Ενημέρωση του πολίτε. Πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες η ενδυνάμωση των πολιτών. Πρέπει να ενισχυθούν. Και αυτό έχει να κάνει και με τις διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν αναφέρεται ουσιαστικά στο έγγραφο η πτυχή αυτή. Και θα έπρεπε να υπάρχει. Μιλάμε για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, μιλούμε για την ανάπτυξη των υποδομών, τις μεταφορές κτλ. Αλλά δεν γίνεται ούτε κουβέντα για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτύου. Ναι, παρακαλώ. Ευρυζωνικότητα, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Πολύ λίγα, πολύ λίγα. Εγώ θα ήθελα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Επίσης παρότερες ενθάρρυνση των πολιτών και καλύτερη ενημέρωσή τους. Όταν μιλάμε για πολύ μικρή συμμετοχή σε όλες αυτές τις διασυνοριακές δραστηριότητες, εμπόριο, υπηρεσίες κτλ. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιήσουν, πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση και συνήθως αυτό που βρίσκουν μπροστά τους μόνο εμπόδια είναι. Τουλάχιστον λοιπόν στο σκέλος στο οποίο εγώ θα είμαι γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο και να ασκήσουμε πίεση για αυτές τις πτυχές. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους ότι η ευρωπαϊκή αγορά βασίζεται στις δυνάμεις της αγοράς. Οι πολίτες χρειάζονται υπηρεσίες και προϊόντα στις κατά το δυνατόν πιο προσιτές τιμές. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν πολύ μεγάλη ενθάρρυνση για καινοτομία, ανταγωνισμό, διασυνοριακές επαφές ένα άνοιγμα εν γέννη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε αυτή την πράξη, την ενιαία αγορά, μέσα σε ένα χρόνο, από, όπως προτείνει ο Επίτροπος ε, Μπαρνιέ, ώστε να μπορέσουμε να δούμε αν τα αποτελέσματα του έργου μας ε, θα είναι απτά. Το είπε και ο Μπαρνιέ. Δεν είναι η βίβλος. Εγώ πάντοτε ανησυχώ λίγο μήπως καταθέσουμε πολλές τροπολογίες και μήπως αυτό το έγγραφο με τις δικές μας εκθέσεις θα είναι κάτι το οποίο θα ισχύει δινικές για την ε, αγωνία αγορά. Όχι, είναι ε, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για τη βίβλο όπως είπα. Τώρα σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομίζω ότι είναι επαρκή διαδικασία. Αντιθέτω, είναι ανεπαρκέστατη και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και αυτό είναι και πρόκληση για εμά, για του ευρωβουλευτέ. Πρέπει να έχουμε επαφέ με του πολίτε, να του ενημερώσουμε, να του ενθαρρύνουμε να ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τις πληροφορίες, για την ενημέρωση. Όλο αυτό το επιπλέον έργο λοιπόν και οι προκλήσεις ουσιαστικά ε, έχουν να κάνουν, είναι για μας γιατί είμαστε οι αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών μας, περιφέρειας μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τούμ. Κύριος Ρέπο λοιπόν. Arvoisa puheenjohtaja, vain muutama yleinen näkökohta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Καρνέτα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και στην παρουσίασή της πολύ καλά μας παρουσίασε τις διαφορετικές διαστάσεις του θέματος. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε την σημασία της ορθής διακυβέρνησης, ε, του του πρέπει να έχουμε διάλογο αποτελεσματικό και αποτελεσματικές εταιρικέ σχέσεις καθώς και αξιολόγηση. Αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι η διακυβέρνηση θα μεταφράζεται και σε πράξη. Ως προς την ίδια την υλοποίηση τώρα αυτών των νομοθετικών προτάσεων στα διάφορα κρατημέλη δεν θα πρέπει να προκύψουν διαφορές στον χειρισμό των ίδιων ζητημάτων από το ένα κράτος στο άλλο. Θα πρέπει να μπορούν οι μεν και οι δε να προχωρήσουν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στα διάφορα κατημέλη με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλες τις εταιρείε και για όλους τους πολίτες. Όπως πολύ σωστά είπε και ο καθηγητής Κορέι Αντεκάμπους, το σημαντικό εδώ είναι η πράξη. Πώς όλα αυτά γίνονται αντιληπτά και ε, εφαρμόζονται στην πράξη. Η ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στην ε, μητρική γλώσσα των χρηστών, των ενδιαφερομένων και τα δίκτυα που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες να λειτουργούν ε, εύρυθμα. εύρυθμα όπως πριν από λίγο είπε και ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ripo. Next, then was... Ευχαριστούμε. Α. Η κυρία Τούμη. Εκ μέρους των Πρασίνων θα είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Ε, δεν ε, είναι βέβαιο ακόμη σε αυτή την φάση της πρώτης ανταλλαγής απόψεων. Όμως νομίζω, όπως σωστά ήδη αναφέρθηκε, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να καταλάβουν ποια είναι τα ενδεχόμενα ωφέλη από την ενιαία αγορά και όχι μόνο να τα καταλάβουν, αλλά να τα αισθανθούν κιόλα στην καθημερινή του ζωή. Δηλαδή, εδώ νομίζω ότι συμμεριζόμαστε όλοι ποιο είναι ο κοινό μα στόχο. Βλέπω να υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα σημεία σε αυτό το κεφάλαιο, όπω για παράδειγμα η πρόταση 26 για ένα κοινό δίκτυο μεταφορών στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό αν θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό πτήσεων εσωτερικώ και να έχουμε ένα δίκτυο υψηλή ταχύτητα στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι μια τεράστια βελτίωση. Επίση, στο 27 για την ενέργεια και τι υποδομέ. Και αυτό είναι ζωτική σημασία για γίνει η βιώσιμη ενέργεια και πιο αποτελεσματική ως προς το κόστος, δηλαδή λιγότερο ακριβή. Και προκειμένου να υπάρξει και μια, ένας υγιής ανταγωνισμός με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Το 29 και το 30 επίσης. Σημαντικά σημεία και αυτά. Διασφαλίζεται η σωστή ισορροπία μεταξύ αγοράς και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ μετά από την υπόθεση... Δεν το κατάλαβα την υπόθεση, μια σχετική υπόθεση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να αναζητήσουμε την ε, σωστή υπηρεσία, ε, τη σωστή ισορροπία. Πρέπει να βρούμε εδώ την κατάλληλη λύση. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των ε, μισθών και των ε, κοινωνικών προτύπων. Διότι αν δεν το πετύχουμε αυτό θα χάσουμε τη στήριξη των πολιτών και των εργαζομένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα λοιπόν αυτό είναι ζωτική σημασία. Και λίγα λόγια για το πρώτο κεφάλαιο, την ε, εσωτερική αγορά των εταιριών. Ε, η Πασκάλ νομίζω θα αναλάβει εδώ. Ο Πασκάλ μάλλον, δεν είναι εδώ σήμερα. Θα τα αναπτύξει και εκείνος ούτως ή άλλως, αλλά εγώ θέλω να τονίσω δύο σημεία να δώσω έμφαση σε κάτι που προτείνει η Επιτροπή το 10 και το 11 για το οικολογικό αποτύπωμα και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Εδώ θα υπάρχει ένας τεράστιος, ένα τεράστιο πεδίο για ανταγωνισμό στο μέλλον. Υπάρχουν δυνατότητες για πάρα πολύ μεγάλες εξοικονομήσεις. Αν μιλάμε για ανταγωνισμό διεθνώ αλλά και εσωτερικός. Πολλά κονδύλια μπορεί να εξοικονομηθούν και κάτι καλό να γίνει και για το κλίμα. Εάν μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά πράσινη επανάσταση στην παραγωγή και την οικονομία μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ωστόσο ότι ο κύριος Κρέσμαν ανέφερε σωστά κάτι σημαντικό εκ μέρους του κυρίου Μπούσο για την καινοτομία. Νομίζω ότι το, το τμήμα που αφορά την καινοτομία δεν είναι ακόμη τόσο σωστά παρουσιασμένο. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε ε, για πάντα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην ε, καινοτομία, αν θέλουμε να ξεφύγουμε και να προχωρήσουμε. Και αυτό πρέπει να τονιστεί εδώ. Πρέπει να επισημάνουμε πού μπορούμε να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πορεία στις επιστήμες, στην έρευνα και το καθεξής. Εδώ νομίζω μπορούμε κάτι να προσθέσουμε στην υπάρχουσα πρόταση. Για τα ευρωμόλογα και αυτό είναι ε, ενδιαφέρον για την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ακόμη, αλλά πραγματικά ε, ανυπομονώ να ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση. Και κάτι που πρέπει επίσης να αναφέρω είναι ότι η Δανία θα προεδρεύει το 2012 όχι με το το δικό μου κόμμα ακόμα δεν είναι κυβερνών κόμμα, όμω το χρόνο έχουμε εκλογέ. Οι πάντε είναι έτοιμοι στη Δανία, άσχετα με ποιο θα αναλάβει την κυβέρνηση τελικά ή όχι. Είμαστε πανέτοιμοι να εργαστούμε για το θέμα αυτό και υπάρχει ε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια πρώτη προτεραιότητα για μας από πλευρά Δανική Προεδρία. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα καλό στοιχείο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενθουσιώδη απάντησή σα και συμφωνώ μαζί σα ε, για την δέσμευση τη Δανική Προεδρία, γιατί ήδη με επισκέφτηκαν υπουργοί από τη Δανία για να προετοιμάσουν την Προεδρία του και αυτό πράγματι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Κύριε Μακλάκ, επόμενη. Ευχαριστώ όλους τους συζητητές για αυτά που είπαν. Εγώ συμφωνώ ότι η ενιαία αγορά είναι το σημαντικότερο, για μένα τουλάχιστον, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πραγματικά ε, πρέπει να προσφέρουμε κάτι στους Ευρωπαίους πολίτες. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να επιτύχουμε το σύνολο, τη μεταφορά του συνόλου της Ευρωπαϊκής Μοθεσία ε, στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση τουλάχιστον για τις ε, θέσεις απασχόλησης. Το κλειδί εδώ είναι μια διαδικασία αμφίδρομης αξιολόγησης, κάτι που έχει προταθεί από την Κομισιόν, το χαιρέτησαν τα κράτη-μέλη. Ε, κάθε στιγμή δεν πρέπει μόνο να ελέγχουμε, να αξιολογούμε, αλλά και να ακούμε και να αντιδρούμε. Αυτό φορά όλους τους εμπλεκόμενους και πάλι για μένα σημαντικό εδώ είναι να συμπεριληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις συζητήσεις για την ενιαία αγορά. Πρέπει λοιπόν να άρουμε όλα τα εμπόδια για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έτσι ώστε να προσφέρουμε πραγματική ε, προστιθέμενη αξία στους πολίτες. Αναφέρθηκε αυτό από την Προραλίσσα, αλλά θα το πω και εγώ. Η ε, ευρυζωνικότητα είναι απόλυτη προτεραιότητα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ενισχύσουμε το πόσο σημαντικό είναι να σημειώσουμε πρόοδο στην ψηφιακή ατζέντα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακλάκεν, λέει ο πρόεδρος. Ίσως εγώ να μιλήσω αργότερα γιατί είμαι και εγώ σκιώδης, εισηγητής. Θα ήθελα τώρα να περάσω σε άλλους ομιλητές ε, κυρία Λούλα μίλησε, Στάιλερ Μανιού μίλησαν, ε, ίσως ε, να κάνω κι εγώ αργότερα κάποια σχόλια. Κοιτάξτε, κι εγώ είμαι σκιώδη συγκήτρια, λέει η κυρία Ρούλε, για το τρίτο θέμα όμως, για την διακυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την κυρία Κανιέτε. Αυτά τα οποία μας είπε εγώ τα στηρίζω ανεπιφύλακτα. Θα ήθελα βέβαια να μου επιτρέψετε να αναφέρω και εγώ ορισμένα θέματα που είναι σημαντικά κατά την κρίση μου. Καταρχήν, όσον αφορά την ε, επέκταση την διεύρυνση του πλαισίου για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, έχουν δείξει οι έρευνες ότι υπάρχουν εμπόδια, ότι υπάρχουν φόβοι στον τομέα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν αρκεί να πούμε επιθυμούμε μόνο τη διεύρυνση, πρέπει να δούμε και πού βρίσκονται τα εμπόδια και πώς είναι δυνατόν να αρθούν τα εμπόδια αυτά, να ε, εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη, να ωφεληθούν όλοι, να είναι πραγματικά ένα βήμα προς τα εμπρός. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε νέα εμπόδια. Η δική μου λοιπόν η εμπειρία με αυτή την αμφίπλευρη ε, αξιολόγηση στην οδηγία υπηρεσιών, η εμπειρία μου ποικίλει. Υπάρχουν δηλαδή κράτη-μέλη τα οποία υπερέβαλαν στην εφαρμογή και αυτό προκάλεσε μεγαλύτερη ε, γραφειοκρατία γιατί εκεί αξιολογήθηκαν και πράγματα που δεν έχουν μεγάλη σημασία. Αυτό λοιπόν πρέπει να διευκρινιστεί. Θεωρώ ότι για τα εργαλεία αυτά πρέπει να επιδιώξουμε τη μεγαλύτερη αποδοχή και τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Και περνάω στο δεύτερο θέμα, στι διαβουλεύσει. Γιατί πριν από την εκπόνηση νομοθεσία ε, έχουμε τι διαβουλεύσει. Θεωρώ ότι τώρα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία για πρώτη φορά με την ε, πράξη περί ενέα αγορά να δούμε πόσο σημαντικέ είναι οι διαβουλεύσει. Κατά πόσο πραγματικά είναι το εργαλείο εκείνο ε, το οποίο μπορεί να κριθεί αποτελεσματικό. Εγώ είμαι τόσο σίγουρη και εδώ αναφέρομαι σε αυτά που είπε η κυρία Τούνεν. Δηλαδή, πιστεύω ότι πάρα πολλές διαβουλεύσεις γίνονται ε, τύπης, ε, γίνονται μέσα από multiple choice ε, έντυπα. Πολλές φορές υπάρχουν και προβλήματα στη γραπτή μετάφραση σε διάφορες γλώσσες και κατά την άποψή μου και η αξιολόγηση δεν είναι η απαιτούμενοι. Άρα δηλαδή όσον αφορά τις διαβουλεύσεις ε, η διαφάνεια υπολείπεται τουλάχιστον για μας, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορούμε να καταλήξουμε κατά πόσον η διαβούλευση απέφερε το ε, προσδοκόμενο αποτέλεσμα ή όχι. Κατά την άποψή μου εδώ πρέπει να επικρατήσει διαφάνεια. Υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά. Να πω και κάτι σχετικά με τις εναλλακτικέ μεθόδους ε, διευθέτησης διενέξεων για τη διαιτησία κυρίως στον χρηματοψηφιακό τομέα, αυτό που προτείνει ο κύριος Μπαρνιέ. Νομίζω αυτό ε, πρέπει να συσχετιστεί και με το θέμα των collective redress, ε, αν θέλετε των ε, συλλογικών προσφυγών για αποζημίωση. Ε, στο Κοινοβούλιο είχαμε μία επιτροπή ε, για το Equitable Life πολύ πριν από την χρηματοπιστική κρίση και κατέδειξε η έρευνα αυτή ότι στον χρηματοπιστωτικό τομέα δεν αρκούν οι εναλλακτικέ μέθοδοι διευθέτησης διαφορών. Ε, πρέπει να υπάρξουν και άλλες για να εμπνεύσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Και κατόπιν, α, μισό λεπτό, χαιρετίζω βέβαια αυτά που είπε η κυρία Κανιάτε σχετικά με το θέμα της ε, στήριξης των μονοαποθυντικών θηρίδων, των one-stop shops. Να έχουμε τέτοιου είδου ε, θηρίδες και το κάνουμε αυτό. Εκ των υστέρων όμως δυστυχώς πολλές φορές δεν προβληματιζόμαστε για τη συνεργασία ανάμεσα σε αυτές τις ε, θηρίδες. Δηλαδή τι κάνουμε, δημιουργούμε άλλη μια ε, διοικητική βαθμίδα, γραφειοκρατία αν θέλετε, χωρίς να προβληματιστούμε από αυτής. Τέλος, όσον αφορά τις παραβάσεις στην έκθεση, το infringement, θεωρώ ότι και εκεί πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, το χρονοδιάγραμμα για τις ε, παραβάσεις, για την ε, ε, διευθέτησή τους, ο φάκελος δηλαδή, πρέπει να ολοκληρώνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Για μένα, ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό είναι οι συμβάσεις οι δημόσιες συμβάσεις. Πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, να τους προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες. Γι' αυτό λοιπόν αυτό, αυτή την πράσινη βίβλο για τις ε, ηλεκτρονικές ε, δημόσιες συμβάσεις, αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον βέβαια γίνεται σωστή χρήση αυτής της δυνατότητας και να έχουμε και ένα συσχετισμό ανάμεσα σε κοινοτομίες και δημόσιες συμβάσεις. Αυτό είναι σημαντικό παράλληλα με το πρόγραμμα πλαίσιο οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορούν και αυτές να αποφεληθούν περισσότερα από τις καινοτομίες. Επ' αυτού ε, πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Και ένα άλλο θέμα όπου δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη με τις προτάσεις του κυρίου Μπαρνιέ είναι για μένα μια ε, χαρακτηριστική περίπτωση για κακές διαβουλεύσεις. Αναφέρομαι στην ε, παροχή υπηρεσιών, στις παραχωρήσεις ε, το να προτείνουμε κάτι πριν έχει ολοκληρωθεί και αξιολογηθεί μία διαβούλευση πριν τελικά όλοι οι εμπλοκόμενοι να τοποθετηθούν θετικά, γιατί όλοι αρνητικοί ήταν, εγώ δεν ξέρω κανείς να μίλησε θετικά για αυτό το σχέδιο, ε, αυτό το βρίσκω πρόβλημα. Γιατί κατά την άποψή μου, όταν ξεκινάει μια διαβούλευση, θα πρέπει να ολοκληρώνεται και να αξιολογείται πριν γίνεται το επόμενο βήμα που είναι να ε, θεσπιστούν νομοθετικές διατάξεις. Ευχαριστώ. Συμφωνώ πλήρω ε, με αυτό που είπατε, ε, ιδίω σε σχέση με τι δημόσιε συμβάσει και νομίζω ότι θα χρειαστούμε και τη δική σα εμπειρία. Θα πω και περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Ολοκληρώνοντα τον κατάλογο, η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ πολύ, Μάλκομ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να μιλήσω για την πρώτη παρουσίαση, αυτό που έλεγε η κυρία Καλνιέτε για μια ολιστική προσέγγιση που πρέπει να έχουμε. Είπατε επίση για τη νέα παρουσίαση για τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω το εξή Αυτή την εβδομάδα είχαμε από την Βουλή των Κοινοτήτων και από το Westminster το ζήτημα των συντάξεων. Και είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρεται και στην πράξη για, τις, για την ενή αγορά. Και νομίζω ότι εμείς ως πολιτικοί ενδιαφέρομαστε για αυτό το ζήτημα και καλό θα ήταν ίσως και ε, στο δικό μας, το, στη δική μου τη χώρα να ενδιαφερθούν και για τις προτάσεις της δικιάς μας. Ό,τι αφορά το 28ο ε, καθεστώς του NTF regime, δεν καταλαβαίνω τι είναι, δεν το ξέρω. Ε, αν μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει. Επίσης, ό,τι αφορά κανονισμούς και οδηγίες και αυτό που είπατε πρώτα κανονισμοί μετά οδηγίες θα το πρέπει να το εξετάσουμε. Και αυτό, αυτό που είπε και η κυρία Τούρουνεν για την συμπερίληψη ε, της κοινωνικής διάστασης στην ατζέντα είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό. Επίσης αμοιβαία ε, προσόντα και τα λοιπά, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων η κάρτα της νολές κίνηση, βελτίωση της κινητικότητας, να μην είναι κάτι για το οποίο απλά γίνεται λόγος, αλλά για το οποίο γίνονται και έργα. Ή ότι θα πρέπει να έχουν κάποια ε, την έννοια ότι τους ανήκει κατά κάποιο τρόπο, ότι ταυτίζονται οι πολίτες με, την, ε, με το θεματολόγιο αυτό. Ίσως στη δική μας ιστοσελίδα τουλάχιστον ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να ή μπορεί ο κόσμος να βλέπει παρουσιάσεις, έγγραφα, και να μπορεί να δίνει και τις ιδέες του. Νομίζω ότι αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να ανοίξουμε, να διευρύνουμε τη συζήτηση. Στη Σκοτία εμεί έχουμε και ένα γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω μιλήσει με τον υπεύθυνο εκεί, ώστε η ατζέντα αυτή να είναι στο δυνατόν ε, πιο ανοιχτή, στο πλαίσιο και αυτής της διαδικασίας δαβουλέσεων που θα έχουμε. Η πρόσβαση στις πληροφορίες επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα ένα άλλο ερώτημα. Πολύς λόγος γίνεται για την ψυχιακή, τη βιομηχανική ατζέντα κτλ. Εμείς, τουλάχιστον εγώ, έχω την εντύπωση ότι και σε άλλες επιτροπές γίνεται λόγος για όλα αυτά τα θεματολόγια, όλες αυτές τις ατζέντε. Και αυτή η ολιστική προσέγγιση που όλοι θέλουμε, που μάλλον δεν συμβαίνει στην πράξη, δεν ξέρω αν υπάρχει ένα ζήτημα ηγεσία εδώ. Ίσως ο πρόεδρός μας θα μπορούσε να τον αλάβει αυτό, να υπάρξει μια πιο κοινή συνεργασία. Υπάρχουν συνάδελφοι στην Επιτροπή Βιομηχανία που μιλούν για την αβιχομική πολιτική, μιλούν για την καινοτομία, για όλα αυτά τα θέματα και πρέπει και εμεί να συμμετάσχουμε στη συζήτηση αυτή. Και νομίζω ότι θα είναι και πιο ισχυρή θέση του Ευρωκοινοβουλίου εάν υπάρχει η κοινή αυτή προσέγγιση. Τέλος. Μίλησα για το ψηφιακό θεματολόγιο που είναι πολύ σημαντικό. Σημείο 2 για την διανοητική ιδιοκτησία, σημείο 5 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ευρυζωνικότητα κτλ. Κυρία Μακλάρκ νομίζω το είπε. Είναι σημαντικά θέματα για τους Ευρωπαίους πολίτες, για όπου ζουν. στη Σκωτία, τις αγροτικές περιοχές που, αγροτικέ που εκπροσωπώ, έχω ακούσει διάφορα. Παραδείγματο χάρη σε μια περιοχή όταν υπάρχει άμποτη δεν έχουν ίντερνετ. Ε, δηλαδή δεν είναι αστείο αυτό που λέω, είναι σοβαρό. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι αν βελτιωθούν οι υπηρεσίε αυτέ ε, θα βελτιωθεί γενικότερα και η αγορά. Θυμάστε που είχαμε το φόρουμ για την ψηφιακή ατζέντα, πόσο δυναμικό υπάρχει, πόσες δυνατότητες υπάρχουν ιδίως και λάμβοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι είναι ίσως μεγαλύτερη πρόκληση. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, βέβαια. Το θέμα της ηγεσία είναι ένα σημαντικό που θα το αναφέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άκουσα ότι ήταν καλό αγώγος στο θαλασσινό νερό κάποτε, αλλά δεν ήξερα ότι επηρεάζει και το ευρωζωνικό ίντερνετ. Κυρία Βερνιό. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα ελαφρώς, αλλά πρέπει να πω ότι άκουσα τους εισηγητές, τον κύριο Μπουσόη, δεν τον είδαμε βέβαια, αλλά θα συνεργαστούμε ε, και με όλους τους υπόλοιπους ε, εισηγητές. Είναι τρία τα σκέλη αυτής της έννοιας αγοράς, ε, όμως δεν μπορούμε να τα αντιπαραβάλλουμε χωρίς να συγκεντριστούν μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, όπως είπε και η Κατρίνα, να συνεργαστούμε όχι μόνο με τις υπόλοιπες επιτροπές, αυτό είναι αναγκαίο, με την Επιτροπή Απασχόλησης, την Επιτροπή Επιχειρήσεων, για τις κοινοτομίες, την Επιτροπή Βιομηχανίας. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είμαστε στη λογική μιας συνεργασίας συλλογικής. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να λάβει μέρη η επιτροπή και ο Επίτροπο ότι για πρώτη φορά, ακόμη και αν συνειδητοποιήσαμε κάποια πράγματα κάπω καθυστερημένα, τουλάχιστον έχουμε ένα κείμενο επιτέλου επί το οποίο μπορούμε να εργαστούμε. Και όλοι μαζί, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, να επιδιώξουμε κοινού στόχου. Είναι ένα κείμενο πολύ φιλόδοξο είναι πολύ ωραία να έχει κανεί υψηλέ προσδοκίε, αλλά προφανώ δεν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα εντό μια θητεία. Τουλάχιστον όμω μπορούμε να ορίσουμε κάποιε πρώτε κατευθύνσει, κάποιου προσανατολισμού. Τώρα για τι επιχειρήσει και την ανάπτυξη, γιατί είμαι συγγέτρια για την ομάδα μου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, νομίζω είναι πολύ σημαντικά όσα έχουν γραφτεί για την βοήθεια προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η εσωτερική αγορά είναι πραγματικό, είναι αλήθεια μάλλον ότι ω τώρα. Ε, έχει δημιουργηθεί για να ευνοήσει τι ε, εμπορικέ συναλλαγέ, αλλά κυρίω για τι μεγάλε επιχειρήσει, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε ε, πραγματικά είναι εκείνε που βρίσκονται πιο κοντά στου πολίτε, πιο κοντά στου καταναλωτέ. Εκείνε δεν έχουν ωφεληθεί καθόλου. Θα έλεγα μάλιστα ότι έχουν δυσκολευτεί από την εσωτερική αγορά. Άρα λοιπόν οι προτάσει που περιέχει το κείμενο αυτό, ιδιαίτερω η εναρμόνιση των εισαγωγικών ε, και κυρίως ο συντονισμός ε, της φορολογικής ε, μεταχείρισης είναι κάτι που μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, ελπίζω ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα καταφέρει να μπορέσει να μετατοπίσει, να επηρεάσει το Συμβούλιο και εδώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρυστεχνία, ιδίω στον τομέα τη ευρωπαϊκή έρευνα, είπαμε προηγουμένω, για το πρόγραμμα πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συνεργαστούμε επί του στόχου αυτού. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε επιτέλου να έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρυστεχνία για τι επιχειρήσει και την ανάπτυξη. Ε, εφόσον βρισκόμαστε στο τομέα των επιχειρήσεων, θεωρώ ότι σημαντικό είναι επίση, και εδώ μιλάμε για εργατικό δίκαιο, μιλάμε για δικαιώματα των πολιτών, είναι σημαντικό λοιπόν και για τις επιχειρήσεις να υπάρχει κάποια μνήμα στο δικαίωμα των πολιτών που αλλάζουν κράτος. Να, να μπορούν να αναγνωρίζονται τα κοινωνικά τους δικαιώματα και στο νέο κράτος, να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αυτά όλα μου φαίνονται πολύ σημαντικά. Πάντως, και το πρόβλημα των επαγγελματικών προσόντων, αυτό που φύγεται στο κείμενο. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ νομίζω ότι προβλέπει αναθεώρηση της οδηγίας του 2005, η οποία είναι τελείως απερχιωμένη σε σχέση με τις εξελίξεις της αγοράς. Εδώ λοιπόν η κινητικότητα, η επαγγελματική κινητικότητα είναι θεμελιώδου σημασία για μια αγορά εσωτερική, η οποία ακριβώς πρέπει να είναι καινοτόμα. Ε, γιατί σε κάθε χώρα ε, υπάρχει κάτι καινούργιο συνεχώς. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να ε, Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι σημαντικό αυτό που μα ε, περιμένει και θα πρέπει να συνεργαστούμε εδώ με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ε, κάτι ακόμη που το προσδοκούσαμε εδώ και πολύ καιρό, η κοινωνική οικονομία. Εδώ πραγματικά νομίζω ότι το να γνωρίσουμε την κοινωνική οικονομία με, μια ιδιαίτερη, ε, με ένα ιδιαίτερο καθεστώ των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, ε, εδώ θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό σε επίπεδο κοινωνική Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα σε συνδυασμό με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, σε κάθε σχετικό ε, τομέα της κάθε χώρας. Για πρώτη φορά επιτέλους ε, υπάρχει αυτό σε ένα κείμενο. Δεν λέω ότι είναι μόνο καλά τα στοιχεία του κειμένου, υπάρχουν και ανακρίβειες, Εδώ πρέπει να εμπαθύνουμε ε, στη συζήτησή μας για την κοινοτομία, λόγου χάρη. Πολύ σωστά η κυρία Τουρούνεν και η κυρία Ριούλε μίλησαν για την πράσινη ανάπτυξη, για τι δημόσιες προμήθειε. Πολύ σωστά η κυρία Ρούιλε μίλησε για του διαγωνισμού εδώ. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και να το δούμε αυτό το θέμα. Πρέπει να ε, προβλέψουμε κοινωνικά κριτήρια, περιβαλλοντικά κριτήρια και να δημιουργήσουμε πραγματικά αγορέ ε, που να επιτρέπουν την πράσινη ανάπτυξη, θέσει απασχόληση, να δώσουν δυναμικό χαρακτήρα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όμω, ταυτόχρονα, Διαφωνώ ελαφρώ μαζί σα. Διότι βρεθήκαμε μαζί σε μια διάλεξη για τι ευρωπαϊκέ μεταφορέ. Και εκεί εγώ συζήτησα τα θέματα αυτά. Η Γαλλία και η Γερμανία ε, επιφυλάσσονται κάπω. Είναι καχύποπτε. Όμω οι υπόλοιπε χώρε είναι πολύ ανοιχτέ στη συζήτηση μια ε, βελτίωση και μεταρρύθμιση ε, προκειμένου να βρεθεί τελικά μια ισορροπία βεβαίω των ε, πρωτοβολιών ε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και του συνδυασμού των δημόσιων ε, υπηρεσιών και των ιδιωτικών. Έχουμε στην Γαλλία τον νόμο ΣΑΠΑ που λειτουργεί πολύ καλά. Σε άλλε χώρε όχι το ίδιο όμω. να βελτιωθούν τα πράγματα και να προχωρήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα κείμενο. Όχι να πάμε σε λάθο κατεύθυνση βεβαίω. Θα προσέξουμε πάρα πολύ. Αλλά εάν θέλουμε να υπάρξει κείμενο πρόταση δηλαδή, ελπίζω εγώ όπως και εσείς ότι θα υπάρξει, ε, θα πρέπει να υπάρξει πρώτα προσεκτική μελέτη, διαβουλεύσει και να λάβουμε υπόψη και τι μέρημνε των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων και των ε, φορέων τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, που είναι οι κατεξοχήν συμμετέχοντες σε αυτές τις εταιρικές σχέσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τι επιχειρήσει πραγματικά σημαντικό για τι επιχειρήσει. Η απασχόληση και η ανάπτυξη πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την καταπολέμηση τη παραποίηση. Είτε μιλάμε για παραποίηση και απομίμηση οποιοδήποτε προϊόντο κυκλοφορεί και μπορεί κανεί να το πιάσει. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζει και βλέπει, αλλά και από το διαδίκτυο. Εδώ πραγματικά έχουμε όλοι το ίδιο πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επινοήσουμε τελείω νέε λύσει. Μιλάμε για μια πραγματική μάστιγα, μια πραγματική καταστροφή που πλήττει την εσωτερική αγορά. Εδώ βρήκα κάτι που ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη ε, στο κείμενο αυτό. Όμως δεν πάει όσο μακριά θα μπορούσε. Διαφάνεια των τραπεζικών δαπανών. Νομίζω ότι είναι καλό να το συζητάμε, μεν, αλλά, και αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές, κατά κύριο λόγο, ε, όταν βλέπουμε την αυτορύθμιση για τις τράπεζες να αναφέρεται, ή την, ε, να δικυβέρνηση. Εδώ ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και είναι πολύ επικίνδυνο όρο, όχι μόνο για του ε, πολίτε και του καταναλωτέ, αλλά και για του χρήστε των τραπεζικών υπηρεσιών, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε πρέπει να προστατευτούν και οι οποίε συχνά πέφτουν θύματα. Θύματα των ε, υπέρογκων τραπεζικών δαπανών. Και δεν έχω πάρα πολλά ακόμη να πω, αλλά φοβάμαι ότι μακρηγόρησα. Λυπούμε. Λυπούμε, και αυτό το ξέρει ο Επίτροπο Μπαρνιέ, το, το λέω εδώ και καιρό, λυπούμε που δεν υπάρχει παρά μία απλή ανακοίνωση για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Λυπούμε ιδιαίτερος που δεν υπάρχει κείμενο, ένα κεφαλαιόδες κείμενο για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Διότι η αγορά μας, η ευρωπαϊκή αγορά, λειτουργεί βάσει μεγάλων επιχειρήσεων, μικρομεσαίων, με πολίτες και καταναλωτές. Όμως επίσης εργάζεται με υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Όλα αυτά είναι υπαρκτά στοιχεία. Εάν θέλουμε λοιπόν αγορά που να λειτουργεί αρμονικά, με δυναμικό χαρακτήρα και, και σε θέση να βρεθεί στο προσκήνιο παγκοσμίω έναντι της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες ε, διαφανείς, ξεκάθαροι, που να γίνονται αποδεκτέ από 27 χώρες και ε, στο εσωτερικό της Ευρώπης να δώσουν δυναμικό χαρακτήρα στην αγορά αλλά και διεθνώ. Μου φαίνεται πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν κάποιε πρώτε ιδέε στο κείμενο, αλλά χρειάζονται διευκρινήσει. Παρά τα καλά στοιχεία πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι θετικά αυτά που λέω, τίποτε δεν είναι τέλειο, όλα χρειάζονται βελτίωση, ακόμα και εμεί οι ίδιοι. Ελπίζω λοιπόν ότι θα εργαστούμε καλά. Ε, για εμά εδώ δεν αμφιβάλλω. Οι τρει εισηγητέ και οι σκιώδε θα συνεργαστούμε αρμονικά, αλλά και η Επιτροπή Ήτρα και η Επιτροπή Απασχόληση και η Επιτροπή Μάλλον και η διάσταση των γυναικών στην εσωτερική αγορά. Μην το ξεχνάμε, η ισότητα των φύλων. Είναι πολύ σημαντικό. Ο επαγγελματικό βίο, ο κοινωνικό βίο. Νομίζω ότι η συνεργασία των τριών αυτών επιτροπών είναι πολύ σημαντική. Βέβαια και με αυτή του εμπορίου. Εννοείται αυτό, είναι αυτονόητο. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό λοιπόν να εκμεταλλευτούμε τι δυνατότητε συνεργασία ώστε να πετύχουμε πριν το τέλο τη θητεία να έχουμε τουλάχιστον αναθέρμανση και να δώσουμε πάλι εμπιστοσύνη στις να προκαλέσουμε την εμπιστοσύνη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή να μπορέσει η Ευρώπη επιτέλου να ανακάμψει και να προχωρήσει σε μια... στο προσκήνιο διεθνώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μπερναντέτ. Πολύ σημαντικά. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπε. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Δεν έχουμε πάει στο δεύτερο γύρο ακόμα. Ο κύριος Κρόιτσμαν δεν έχει μιλήσει ακόμη. Δεν θα δώσω το λόγο σε όσους έχουν ήδη μιλήσει μια φορά. Πρώτα θα δώσω σε αυτούς που δεν έχουν. Κύριο Κρόιτσμαν. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιε παρατηρήσει, γιατί είμαι σκιώδη εισηγητή. Να τοποθετηθώ πάνω σε όλο αυτό το θέμα. Αναφέρθηκε ήδη ε, το ότι για τον καταναλωτή η δημιουργία της ε, ενιαίας αγορά είναι μια τεράστια πρόοδο. Έχει αναφερθεί επανειλημμένα ότι δεν πρέπει να έχουμε μόνο κατά νου τις επιχειρήσεις αλλά και τους ε, καταναλωτές. Εδώ λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να προκαλέσουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αυτό είναι καλό, πάντα καλό. Καλύτερα να υπάρχει ανταγωνισμός από το να υπάρχουν ε, μονοπωλιακές ε, τιμές. Αυτό το βιώνουμε στη Γερμανία. Εκεί δεν έχουμε μονοπόλια αλλά έχουμε ολιγοπόλια. Και διαπιστώνουμε ότι τα Σαββατοκύριακα παραδείγματο χάρη, ανεβαίνουν οι τιμέ βενζίνη. Ε, κατά κάποιο τρόπο γίνεται αυτό συντονισμένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ορισμένε επιχειρήσει να μπορούν να αποκλίνουν. Τώρα, όσον αφορά το ε, ψηφιακό μέρισμα, νομίζω και αυτό θα ωφελήσει τον πολίτη στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε. Το τρίτο θέμα, σημαντικό για τους πολίτες, είναι η αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ε, την ενιαγορά αγορά μπορούμε να τη φέρουμε πολύ κοντά στους πολίτες ε, διότι είναι απαραίτητο να υπάρχει κινητικότητα. Εχθές ε, είδα σε μία σε ένα φιλμ τσέχους γιατρούς ε, που κερδίζουν 1000 ευρώ και αυτοί παρετήθηκαν από τη δουλειά τους για να πάνε να εργαστούν στη Γερμανία ή στην Αγγλία που μπορούν να κερδίσουν πολλά περισσότερα χρήματα. Στην ενιαία αγορά λοιπόν υπάρχει κινητικότητα και ως εκ τούτου η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είναι πολύ σημαντική. Όπως επίσης ε, και η ε, δημιουργία μιας επαγγελματικής ταυτότητας. Μια ταυτότητα που θα επιτρέπει το να εργάζεται κανείς διασυνοριακά. Αυτό θα αφορά ενεργούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ε, εποπτείας της αγοράς. Να υπάρχει καλύτερο συντονισμός ε, τα τελωνία και στις άλλες αρχές, όπως και κοινέ κατευθυντήρες γραμμές για τον έλεγχο της ασφάλειας ποιότητας. Αυτό θα είχε δύο ωφέλη. Αφενός, καλύτερη προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα προϊόντα και αφετέρου δημιουργία θεμητού ανταγωνισμού για τους παραγωγούς, οι οποίοι όμως τηρούν τις ε, προϋποθέσεις ασφαλείας. Δεν θα κουραστώ να αναφέρω ότι η εποπτεία της αγοράς στο θέμα αυτό πρέπει κάτι να σκεφτούμε, διότι έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα κάθε χρόνο συμβαίνει το ίδιο. Εμφανίζονται παιχνίδια στην ευρωπαϊκή αγορά που ε, δεν μας ε, εκπροσωπούν. Και οποτεδήποτε γίνεται μια συζήτηση και γίνεται τώρα μια τέτοια που είναι οι αδυναμίες, ε, βλέπουμε ότι ας πούμε τα κινέζικα παιχνίδια έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κέντρο της, μέσα από το Ρότερνταμ. Εάν λοιπόν κατορθώσουμε να αναλάβουμε όλοι από κοινού τις ευθύνες μας. Εγώ έχω προτείνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει η Frontex. Τα κράτη-μέλη είναι αλληλέγγυα με τις χώρες ε, τις ε, παράκτης αν θέλετε που αισθάνονται πρώτες το πρόβλημα των μεταναστών. Εκεί λοιπόν υπάρχει η Frontex. Γιατί να μην υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και στην εποπτεία της αγοράς. Οι επίτροποι οποτεδήποτε τους κάνω μια σχετική ερώτηση μου λένε αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και γνωρίζουμε ότι ε, αν τα κρατημέλη προσέξουν λιγάκι τον, την σωστή επάνδρωση των τελωνιακών αρχών θα αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημα. Πάντως είναι ένα πρόβλημα και εγώ ήθελα να το αναφέρω. Προηγουμένως αναφέρθηκε και κάτι άλλο. Το θέμα των συλλογικών προσφυγών. Οποτεδήποτε συζητιέται κάτι τέτοιο στην Ευρώπη ε, θα πρέπει να το συζητάμε πολύ προσεκτικά. Αφενός ε, έχουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, ε, τα διεκδικούν οι καταναλωτές, πολύ σωστό αυτό. Από την άλλη όμως ε, πρέπει να σας προειδοποιήσω, δεν είναι εύκολο να εφαρμόσουμε εδώ στην Ευρώπη το αμερικανικό δίκαιο. Αυτό δεν θα εξυπηρετήσει ούτε τους καταναλωτές ούτε τις επιχειρήσεις. Να μην το κάνουμε αυτό το λάθος. Πράγματι στο θέμα αυτό πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις, πρέπει να αναλάβουμε ενέργειες και πρέπει να συζητήσουμε. Τέλος, ε, ο κατάλογος των μέτρων δεν είναι πλήρης. Παραδείγματο χάρη, δεν αναφέρονται τα τέλη περιαγωγής, ότι αυτά πρέπει να καταργηθούν μέσα το 2015. Δεν αναφέρεται αυτό το μέτρο. Ε, γίνονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις, μικρό το χρονικό περιθώριο. Ε, είμαι σίγουρος όμως ότι κάτι θα γίνει. Και κάτι άλλο που αναφέρθηκε προηγουμένως, πρέπει να ε, ταυτιστούμε καλύτερα, να συνεργαστούμε καλύτερα με τις άλλες επιτροπές για να μην υπάρχουν επικαλύψεις στις εργασίες μας. Εμείς εστιάζουμε την προσοχή μας στην ενιαία αγορά, είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να μεριμνήσουμε οποτεδήποτε γίνονται παραμφερείς εργασίες σε άλλες επιτροπές και εκεί να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση της ενιαίας αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, ε, και επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ τις ε, παρατηρήσεις με την ιδιότητά σας ε, του Πρόεδρου της Επιτροπής και ως ε, σκιώδης συγητής της έκθεσης της κυρίας Καρνιέτη. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Καρνιέτη, το τι πρέπει να επιτύχουμε τους επόμενους τέσσερις μήνες. Νομίζω είχε δίκαιο αναφέροντας ότι ο ρόλος κλειδί αυτής της Επιτροπής είναι να ιεραρχήσει τα θέματα και να εντοπίσει τους τομείς εκείνους όπου επιθυμούμε να αναλυθούν ενέργειες για τις 15 προτάσεις. Σε τελική ανάλυση δεν πρόκειται για ένα, μια εναρμονισμένη νομοθετική πρόταση και ούτε ήταν και αυτός ο σκοπός. Πρόκειται για ένα καθαρά πολιτικό έγγραφο με πολύ μεγάλη σημασία. Κύριε Σβάπ, κύριε Σβάπ, με συγχωρείτε, απευθύνομαι στην Επιτροπή αν θέλετε να μιλήσετε στον συνάδελφό σα ε, να το πράξετε αυτό εκτό τη αίθουσα. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα επικοδομητικό ε, αν όλοι οι συγητέ και οι σκιώδει συγητέ εστιάζανε την προσοχή του στο πολιτικό μήνυμα που θέλουμε να εκπέμψουμε. Νομίζω λοιπόν από τι συζητήσει που έχουν γίνει μέχρι τώρα κατέστη σαφέ ότι οι περισσότεροι από εμά, Πρόεδρε διακόπτη πάλι. Κύριε Ρούλε, σα παρακαλώ. Ξέρω ότι υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν για τα ε, δομικά υλικά. Και αυτά μπορείτε να τα συζητήσετε εκτός της Πρόεδρος λοιπόν και πάλι λοιπόν, όσον αφορά την αξία που πρέπει να προσθέσουμε στη διαδικασία, εγώ έχω την άποψη ότι στις ε, περισσότερες περιπτώσεις ε, για τις 15 προτάσεις συνάδελφοι είναι ικανοποιημένοι. Ίσως θέλουν να προσθέσουμε κάτι, ε, αλλά θεωρούν ότι η Κομισιόν έκανε καλή δουλειά. Οι 30 προτάσεις είναι πάρα πολλές για να δώσει κανείς μία κατεύθυνση και μερικά πράγματα επαναλαμβάνονται. Ενώ λοιπόν συμφωνώ με την κυρία ότι ε, όσον αφορά το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη η Επιτροπή δεσμεύτηκε να το αναθεωρήσει. Αυτό ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μια δική μας πρόταση. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κρίσιμη τομής όπου πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κρατη να επιταχύνουν ε, τις διαβουλεύσεις, να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες έτσι ώστε να λειτουργεί καλύτερα η ενιαία αγορά σε πάρα πολλούς τομείς. Ε, νομίζω έχουμε αναφερθεί σε πολλά όπως ε, στην ολοκλήρωση, στην εδραίωση, σε όλους τους τομείς ε, να υπάρχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, γραμμές που προσφέρουν βοήθεια Αυτή τη στιγμή δυσκολεύουμε λιγάκι να εκφραστώ, αλλά όλα αυτά τα θέματα θέλω να πω είναι τομεί όπου τα κράτη-μέλη μπορούν κάλλιστα να προχωρήσουν ταχύτατα. Και όσον αφορά παραδείγματο χάρη την οδηγία υπηρεσιών, εκεί πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη, ήδη επενδύσει πολλά χρήματα για αυτέ τι μόνο απευθυντικέ ε, θηρίδε. Ε, πρέπει λοιπόν όλα αυτά να χρησιμοποιούνται. Κάτι άλλο, κάπω ευρύτερο θέλω να πω. Ε, κάτι που απογοητεύει, στο οποίο απογοητεύει η, ενιαία, η πράξη αυτή περί ενιαίας αγοράς. Ενώ θέλουμε να προβάλλουμε την αξία της ενιαίας αγοράς στους πολίτες, στους επιχειρηματίες και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να τους ενθαρρύνουμε να εμπλακούν περισσότεροι σε αυτή τη διαδικασία. Θα θυμάστε ότι όταν είχαμε την ακρόαση ε, περί της οδηγίας υπηρεσιών υπό την καθοδήγηση της κυρίας Κέπχαρτ, ε, ορισμένες χώρες είπαν ότι παίρνουν περισσότερα ερωτήματα από τις, χώρες, από τις επιχειρήσεις της χώρας τους για δυνατότητες εμπορίου από ότι από επιχειρήσεις εκτός χώρας τους. Πολλοί είπαν ότι οι πολίτες δεν βλέπουν τα πλεονεκτήματα. Οι πολίτες ε, είναι και αυτοί μικρές, ε, μεγάλες επιχειρήσεις, ε, είναι εργαζόμενοι οι επιχειρήσει τους εμπλέκονται στην ενιαία αγορά και ίσω να μην βλέπουν απαραίτητα όλες αυτές τις διασυνδέσεις. Όμως πιστεύω ότι εκεί όπου πραγματικά απογοητεύονται οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις γιατί πιστεύουν ότι η νέα αγορά δεν τους προσφέρει πολλά πράγματα και αν εκείνες δεν το αισθάνονται τότε προφανώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό ω προ την αποδοτικότητά μα. Ορισμένα λοιπόν θέματα που δείξατε κι εσεί, αλλά κυρίω η Ρία Ρούλε, δηλαδή την δυνατότητα πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, αυτό είναι κάτι που τα κράτη-μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι στου κανονισμού που να του εμποδίζει, αλλά ο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται οι ε, κανονισμοί, αυτό είναι αποτρεπτικό. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία ε, Κανιατέ για την διακυβέρνηση. Το θέμα των δημόσιων συμβάσεων είναι καθοριστική σημασία. Εκεί μπορούμε να προσθέσουμε αξία, όπω ήδη το πράξαμε. Υπάρχουν τομεί όπου υπάρχουν δημόσιες συμβάσεις ε, για να προωθηθούν οι πράσινε ε, συμβάσεις Ξέρουμε λοιπόν ότι δεν απαραίτητο να πράξουν τεράστιε αλλαγέ στο νομικό πλαίσιο. Η Κομισιόν θα το ελέγξει αυτό, αλλά εκεί παραδείγματο χάρη αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Είναι θέμα ερμηνεία, παρουσίαση, εκπαίδευση, πρόκληση δραστηριοτήτων και ε, ένα μέρο του προβλήματο είναι ότι οι δημόσιε συμβάσει δεν αντιμετωπίζονται ω ένα εργαλείο τη ενιαία αγορά έτσι ώστε να υπάρχει ε, καλύτερο ανταγωνισμό για τι δημόσιε συμβάσει, τι ε, πράσινε συμβάσει και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, στη Σουηδία, παραδείγματο χάρη, κατά διάρκεια τη Σουηδική Προεδρίας, θα θυμάστε, αναφέρθηκε στη χώρα αυτή οι δημόσιε συμβάσει και η εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία εμπίπτουν σε αρμοδιότητε τη αρχή ανταγωνισμού τη ε, Σουηδία, γιατί επιθυμούν να έχουν μια δίκαιη και ανοιχτή αγορά. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τομεί που μπορούμε να προσθέσουμε αξία. Αυτό που κατ' ουσίαν λέω είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε τα εργαλεία την πλατφόρμα, θα θυμάστε τη λέξη που χρησιμοποιήσε ο κύριος Μόντι, την πλατφόρμα λοιπόν, ε, πάνω στην οποία μπορούν να προσφερθούν και άλλες πρωτοβουλίες. Και συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε αρκετοί από εσά για την πολιτική καινοτομία, στη βιομηχανική πολιτική ε, στον 21ο αιώνα. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να επαναλαμβάνουμε πράγματα εκεί όπου ήδη έχουμε αναλάβει ευθύνες. Ε, η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει Ας πούμε, ε, όσον αφορά την Ένωση Καινοτομίας, ε, κατέστη σαφέ ότι εκεί οι ε, συνάδελφος είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι ως προς την κινητικότητα των ερευνητών και θέλει αυτό να το χρησιμοποιήσει ως τη λιβύα Λίθο για να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή συνεργασία γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν πραγματικοί περιορισμοί στην έρευνα στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε συλλογματικά. Μπορούμε να επιλέξουμε τέτοιου θέματα, να τα προβάλλουμε και το τελευταίο το οποίο θέλω να αναφέρω αφορά στη διαδικασία. Γιατί πολλοί από εσά αναφερθήκατε στο πόσο σημαντικό είναι να εμπλακούν και άλλε επιτροπέ. Είχαμε ενθάρρυνση και ενθαρρυντική απάντηση από άλλε επιτροπέ. Τι κάλεσα εγώ να στείλουν τι εκθέσει του. Μερικέ το έπραξαν αμελητοί. Ε, βέβαια, ε, είπα να γίνουν όλα αυτά ανοιχτά και ένα από τα πράγματα, πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνουν να δημοσιεύσουμε εμείς το δικό μας το χρονοδιάγραμμα για την ανταλλαγή απόψεων. Να δούμε κατά πόσον μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις άλλες επιτροπές που εργάζονται επί του θέματος να ε, συναντηθούν με τους δικούς μας εισηγητές. Νομίζω η συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί κατέδειξε ότι οι εισηγητές είναι πρόθυμοι να εξετάσουν το θέμα σε τρεις εκθέσεις. Ε, το γεγονός λοιπόν ότι ε, περιλαμβάνουμε πάρα πολλούς ανθρώπους από ένα μεγάλο πολιτικό φάσμα, αυτό είναι θετικό και ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει τώρα εδώ να διαφωνούμε και να τσακωνόμαστε για τις αρμοδιότητες, δεν χρειάζεται, γιατί το σημαντικό θέμα είναι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η κατανομή ή ανακατανομή των πόρων που υπάρχουν για να προχωρήσουμε. Πρόκειται λοιπόν για μια ευκαιρία, όπως είπατε και εσείς, για να επανέλθει η ενιαία αγορά, κάτι το οποίο είναι και ο στόχος και η φιλοδοξία της έκθεσης Μόντι. Νομίζω ότι πρέπει να τα εξετάσουμε τα θέματα κάτω από το λειτουργικό στοιχείο. Καλό λοιπόν που εμπλέκονται όλοι οι συγητές. Νομίζω και κλείνω πραγματικά λέγοντάς σας Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι επιτύχαμε σημαντικό, είχαμε μεγάλο πολιτικό βάρος. Περάσαμε πολιτικό μήνυμα με την πρώτη έκθεση, γιατί είδαμε ότι όλα τα κόμματα στήριξαν αυτό το μήνυμα. Αν θέλουμε λοιπόν ε, να πούμε στις κυβερνήσεις ότι πραγματικά εδώ χρειαζόμαστε δράση, ε, μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο και με αυτή την έκθεση και οι ε, εκθέσεις πρωτοβουλίας ε, είναι επιτυχημένες μόνο εφόσον έχουν μεγάλη απήχηση. Από τη φύση τους έτσι είναι οι εκθέσεις αυτές. Σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και σίγουρα θα συνεργαστούμε με τον κύριο Ντεκάπος, εγώ θα το πράξω αυτό, στις ε, δικές μου, στο δικό μου τον τομέα δραστηριοτήτων. Ε, υπάρχει βέβαια μετά και μια συνεδρία συντονιστών και θέλω να επενθυμίσω σε όλους σας ότι οι συντονιστές ε, οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη υπό τη δική μου βέβαια την καθοδήγηση. Θα καλέσουμε τους τρεις συγητές να έρθουν στη συνεδρίαση των συντονιστών ο κύριος Μπουζόου δεν είναι πια συντονιστής, ο κύριος Κρόιτσμαν είναι εισηγητής. Θα έρθουν λοιπόν και οι εισηγητές στις συνεδρίες των συντονιστών για να εξετάσουμε την πρόοδο των θεμάτων. Αυτά. Εκείνο που θέλω να κάνω είναι Βλέπω ότι είναι εδώ κύριε Μπράμπτον με μια δυνατή ομάδα από την Κομισιόν και θα ήθελα να τη ρωτήσω μήπως και εκείνη θέλει να κάνει κάποια σχόλια, να μας πει ε, πώς θα προχωρήσει κατά την άποψή μας η διαδικασία διαβουλεύσεων. Ε, και κατόπιν βέβαια θα έχουμε και τα ε, καταληκτικά σχόλια από τους τρεις εισηγητές ε, ίσως αν θέλει να μιλήσει και ο κύριος Σβάμπ. Ε, λοιπόν, πρώτα η Κομισιόν και μετά ε, μπορείτε αν θέλετε να μιλήσετε γιατί θα έχουμε χρόνο μέχρι τις 11.30. Κυρία Μπρόμπτε πρώτα απ' όλα. Μήπως θέλετε εσείς να σχολιάσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, βουλευτές που τοποθετήθηκαν σήμερα το πρωί. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μας η συζήτηση. θεωρούμε και συγκρατούμε ότι υπάρχει ευρεία στήριξη για την γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή την ανακοίνωση και ιδιαίτερος για την ανάγκη να ε, επικεντρωθούμε σε τρεις πυλώνες στο σχεδιασμό των δράσεών μας, δηλαδή για τις επιχειρήσεις, αλλά αποκαθιστώντα και την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών και ξαναβλέποντα την κυβέρνηση τη ενιαία αγορά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ε, ακολουθώντα σε γενικέ γραμμέ αυτή την ε, προσέγγιση. Πρέπει να πω ότι την προσέγγιση αυτή τη στηρίζει και το Συμβούλιο, διότι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα ε, εργάστηκε επί του θέματο αυτού το ανέλαβε δηλαδή αυτό και αύριο ήδη θα συνεδριάσει προκειμένου να εγκριθεί ένα πρώτο σχέδιο συμπρασμάτων ενό στάδιου μεταβατικού, ε, ενδιάμεσου μάλλον. Διότι το Συμβούλιο, ενώ εγκρίνει το ή άλλω την προσέγγιση μα, δεν έχει παρόλα αυτά καθορίσει το ίδιο τι προτεραιότητέ του. Είναι λοιπόν ένα έργο που το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να κάνει ε, και είναι σημαντικό από τη δική μα την Σκοπιά η θεσμικά όργανα σε αυτή την περίοδο που έχουμε ακόμη μπροστά μας να εργαστούν από μια ημερομηνία και μετά, ε, στιγμή που θα ορίσουμε βέβαια ανάλογα με το πώς προχωρήσουν ε, οι συζητήσεις και στο δικό σας επίπεδο, προκειμένου να καταλήξουμε σε ευρεία πολιτική συμφωνία για τις προτεραιότητες που όλοι θέλουμε να προωθήσουμε για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη διαδικασία, κάποια στιγμή που θα οριστεί μελλοντικά, θα πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί, ώστε να δούμε κατά πόσον συγκλίνουμε. Και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν το εγχείρημα αυτό, ώστε να καταλήξουμε σε χειροπιαστά μέτρα, μέτρα τα οποία από ένα σημείο και μετά θα μπορούμε να υλοποιήσουμε, γιατί τα όσα έχουν προβλεφτεί για την ώρα για τη, διακυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη συζήτηση, που δεν μπορώ να την ονομάσω τριμερή διάλογο, όμω πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένα παραλληλισμό με την νομοθετική διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι ζωτική σημασία και θα γίνει μετά το στάδιο των διαβουλεύσεων. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή θα ετοιμάσει μια ανακοίνωση σε συνθήκε πλήρους διαφάνεια και θα πρέπει και θα ληφθεί κάποια απόφαση από τα τρία θεσμικά μας όργανα για τις προτεραιότητές μας. Υπάρχει ένα, μια σειρά ερωτημάτων και ανάλογα με το χρόνο που μας έχει κατανεμηθεί, δεν μπορούμε να τις καλύψουμε όλες τώρα, όμως όπως είπατε, ε, είναι πολύ σημαντικές ε, οι επόμενες κινήσεις μας για το θέμα αυτό. Θα δούμε κατά πόσον και δημερός μπορούμε να απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα ε, υπάρχουν ε, κάποια σημεία που φαίνονται αρκετά δύσκολα να διαλευκανθούν, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια καλή, καλό έκβαση στις συζητήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι θετικό το ότι το εξετάζει και το Συμβούλιο και γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει μια ευθυγράμμιση μεταξύ μας. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον και αυτό που είπατε ότι θα τα λάβει υπόψη η Κομισιόν στην τελική της έκθεση. Πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί. Ξέρετε λοιπόν ότι είναι μια πρόταση ανοιχτή σε διαβουλεύσεις, άρα είναι πολύ σημαντικές οι πολιτικές μας ε, τοποθετήσεις. Πολύ καλά, νομίζω ότι έχουμε χρόνο για να ακούσουμε για δεύτερη φορά τους ε, εισηγητές, αλλά νομίζω ότι και ο κύριος ε, Σφάπ θέλει το λόγο ο κύριος Κρόιτσμαν, ο καθηγητής Κορέα Ντεκάμπος και η Ακαλνιέτ. Πρώτος ο κύριος Σβάπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω το εξή. Βγήκα έξω για λίγο και μίλησα με κάποιον από τους συνεργάτες μου, γιατί δεν είναι δυστυχώς ο κανονικός μου συνεργάτης, ο βασικός μου συνεργάτης εδώ. Πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι είναι εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από όλους, ε, από τους συγητές. Ε, θέλω να τους ε, συγχαρώ και τους τρεις να τους ευχαριστήσω. στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και χρειαζόμαστε βέβαια μια μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποια βάση θα προχωρήσουμε. Και πρέπει να πω ότι είναι σωστό να ακολουθηθεί μια ολιστική προσέγγιση. Φυσικά βέβαια θα πρέπει να δούμε και κάποια συγκεκριμένα αιτήματα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι τα αιτήματα που θα διατυπώσουμε και μετά θα πρέπει να εμείνουμε σε αυτά. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν για το τι θέλουμε να συμπεριληφθεί στις εκθέσεις, θα πρέπει να φροντίσουμε να πάρουμε με το μέρος μας όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές. Υπάρχει το ζήτημα ε, των συλλογικών προσφυγών, που πρέπει να το έχουμε κατά νου, αλλά βέβαια το βασικό ζήτημα, όπως υπόθηκε, είναι η υλοποίηση. Και φοβούμε, αλλά μάλλον θα υπάρξουν και κάποια ζητήματα με την ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο που πολύ σωστά επισήμανε και ο κύριος Κορέντα Ντεκάμπους. ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πολίτες. Και βέβαια πρέπει να συναγάγουμε και κάποια πρακτικά συμπεράσματα. Έχουμε 800 ρυθμιστικούς φορείς. 200 όμως ε, μιλάμε για τομείς συγκεκριμένα, οι 200 τομείς ρυθμίζονται μόνο σε ένα κράτος ε, μέλος, όχι σε περισσότερα του ενός. Θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται τα επαγγέλματα. Αυτό αφορά και τις δημόσιες προμήθειες. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο έτσι όπως έχει κατάσταση ότι η Επιτροπή μας είναι πρόθυμη να καταβάλει προσπάθειες για να υπάρξουν βελτιώσεις εκεί όπου αυτό είναι δυνατό. Η Επιτροπή λέει ότι είναι δυνατό να υπάρξουν βελτιώσεις, αλλά μέχρι να τις δούμε επιτάπητος τις σχετικές προτάσεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θέλω να προσθέσω το εξής. Αν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε την πλειοψηφία πίσω από αυτή την ολιστική προσέγγιση, θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τις άλλες επιτροπές που συμμετέχουν σε αυτή την νομοθετική διαδικασία. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κάποιες φορές το Κοινοβούλιο κατηγορείται ε, για τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Ε, νομίζω ότι το ΑΕΛΚ πρέπει να συνεργαστεί, όλοι πρέπει να συνεργαστούν και για να ολοκληρώσω θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καλνιέτε. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία βέβαια όπου η διακυβέρνηση και μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί. Αναφέρθηκε ένας μηχανισμός για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι στο προσκήνιο των προσπαθειών μας, αλλά και ε, στο προσκήνιο των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη επίσης μας υποστηρίζουν και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να τα έχουμε και αυτά στο πλευρό μας και σίγουρα θέλουμε να υπάρξει συνεργασία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Αντρέα, σε ευχαριστώ που δείχνεις ότι υποστηρίζεις τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές σου για συνεργασία του ΕΛΚ με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Είναι σημαντικό να φτάσουμε σε μια κοινή προσέγγιση έτσι θα μπορέσουν και οι συγητέ να φέρουν σε πέρα σε αυτή την πολύπλοκη δέσμη προτάσεων. Νομίζω ότι η κυρία Βενιώτη, πρόεδρός μου, θέλει να προσθέσει κάτι. Θα τα πω πολύ σύντομα, γιατί αυτό είναι ένα συμπέρασμα. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι έχουμε ένα κείμενο πολύ πλούσιο, ιδιαίτερα φιλόδοξο και συμμερίζομαι απόλυτα αυτό που είπε ο Πρόεδρος. Πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες και πολιτικά μηνύματα. Αυτά που θέλουμε να αποστέλει η εσωτερική αγορά και η πρότασή μας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης όλοι είχαμε περίπου καμιά δεκαριά προτεραιότητες ε, για τις οποίες μπορούμε ήδη να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για να δούμε αποτελέσματα αρκετά σύντομα. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε οι προτεραιότητες αυτές να οριστούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο εφόσον η Επιτροπή μας είπε ότι υπάρχει συνεδρίαση αύριο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα. Ελπίζω λοιπόν ότι οι ήδη θα μπορέσουν και εκείνοι να ορίσουν κάποιε προτεραιότητε από την πλευρά του και να έχουμε την ε, πληροφορία αυτή πολύ σύντομα για να δούμε κατά πόσο συμφωνούμε μαζί του και να έχουμε κι εμεί πρόσβαση στο κείμενο αυτό, κείμενο τη Επιτροπή. Αλλά νομοθέτε είναι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε μαζί για πολλά πράγματα, όχι μόνο με το Κοινοβούλιο, αλλά και με του νομοθέτε μα, το Συμβούλιο. σω εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα γιατί έχουμε 27 χώρε, όμω και το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά πιεστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μπερναντέτ. Ας ε, ακούσουμε τις γρήγορες απαντήσεις και σχόλια των ε, εισηγητών. Ο κύριος ε, Κρόιτσμαν πρώτα. Θέλει να προσθέσει κάτι άλλο, να κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ σύντομο. αυτά που είπε ο κύριος Βάπη είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να προσέξουμε όταν θα έχουμε γκρίνει το κείμενο να ακολουθήσει και η εφαρμογή του στα κράτη-μέλη. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να θεσπίζουμε μια οδηγία ή ένα κανονισμό ή οτιδήποτε και εκ των υστέρων να διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν αυτά τα κείμενα. Τώρα λοιπόν, λόγω της οικονομικής κρίσης, ε, σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύσκολο να ενθουσιάσει κανείς τους πολίτες για την Ευρώπη, όμως ε, αν παρακολουθήσετε λιγάκι τις συζητήσεις ε, που γίνονται αυτές οι μέρες, θα ακούσετε ότι αυτό που λείπει είναι ο ηγέτης, ο που θα προβάλλει την Ευρώπη. Ως εκ τούτου επικρατούν όλο και περισσότερο τα εθνικά συμφέροντα. Άρα δηλαδή ε, οι προτάσεις ε, για τις οποίες ε, συζητάμε και σίγουρα θα τις συμπληρώσουμε γιατί η Κομισιόν έκανε 15 προτάσεις, αλλά θα υπάρξουν ίσως και βελτιώσεις, γιατί πρέπει να υπάρξει ενιαία αγορά και πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς στο ότι οι πολίτες ε, καλό είναι να έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς που εργάζονται για αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, καθηγητής Ντεκάμπος. Πολύ γρήγορα βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση ότι υπάρχει ομοφωνία για διάφορα θέματα. Αυτό δεν ίσχυε πριν από έξι μήνες ή πριν από ένα χρόνο. Ο κύριος Κρόιτσμαν είπε ότι θα πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό είναι πράγματι πάρα πάρα πολύ αναγκαίο. Πολλοί ομιλητές ακριβώς ε, έθεσαν το θέμα αυτό και θα πρέπει το σχέδιο να είναι πραγματικά προσαρμοσμένο στους πολίτες, στα κράτη-μέλη. Και όπως είπε και η Κομισιόν, νομίζω ότι το είπε η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι κυρίαρχα στα σχέδια, αλλά και οι πολίτες θα πρέπει να νιώθουν ότι ταυτίζονται, ότι τους ανήκουν αυτά τα σχέδια. Ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με την ενημέρωση των πολιτών, σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια, όλα αυτά είναι σημαντικά. Σημαντικό επίσης είναι να υπάρχει συντονισμός και με τις άλλες επιτροπές. Μιλήσαμε για πολλά ζητήματα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενημέρωση, όλα αυτά τα θέματα. είναι στο επίκεντρο της ε, ενιαίας αγοράς. Εγώ δυσκολεύομαι κάπως. Ε, ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε την ομοφωνία για τις συλλογικέ προσφυγές, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να εργαστούμε. Δεν είμαι δύσπιστος, δεν είμαι σκεπτικιστής, απλά νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταλήξουμε. η απόφαση για την κατανομή σε τρεις εκθέσεις ήταν ευφυής απόφαση και χρήσιμη. Βέβαια, η διαχείριση αυτών των τρων εκθέσεων θα είναι απαιτητική, θα είναι δύσκολη, αλλά είναι σημαντικό να τα καταφέρουμε. Είναι απαιτητικό το όλο εγχείρημα, αλλά και γιατί το ζήτημα της ενίας αγοράς δεν είναι ένα ζήτημα που προσελκύει, που είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, ως, ε, να, το κάνουμε ελκυστικό και να ε, του δώσουμε την προβολή από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά παρόλα αυτά ε, πρέπει να τα καταφέρουμε. Thank you very much. And then to conclude, Mrs. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Καρνιέτα, για να κλείσουμε. I would like to join all my Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους που μας είπαν ότι όλα αυτά γίνονται για τους πολίτες. Το δικό μου ε, μέρος αφορά το πώς η διακυβέρνηση της εσωτερική αγοράς θα μπορέσει να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη για τους πολίτες. Βεβαίως, με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να πω, ότι το έγγραφο αυτό, η πράξη για την ενιαία αγορά, θα δώσει μεγαλύτερη προβολή στην ενιαία αγορά μεταξύ των προτεραιοτήτων ε, του Κοινοβουλίου συνολικά. Ε, και αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και τους σκεώδεις εισηγητές για την αφοσίωσή τους θέλουν όλοι από ό,τι φαίνεται να καταλήξουμε σε μια έκθεση επικοδομητική που να εγκριθεί με ευρία πλειοψηφία στην Επιτροπή και ελπίζω και στην Ολομέλεια. Επίσης, να πω ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστώ που όλοι όσοι παρενέβησαν σήμερα υπογράμμισαν τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης για αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο. Να απαντήσω στην κυρία Τάιλερ για το καθεστώς TNA. Εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκούς κανόνες που δεν έχουν αντικαταστήσει τους εθνικούς, αλλά είναι εθελούσια η χρήση τους. Είναι μια εναλλακτική λύση. Για παράδειγμα χρησιμοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Καταστατικό εταιρεία. Οι κανονισμοί, οι οδηγίε, τι πρέπει να υπηρεσχύσει. Συμφωνώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί οι κανονισμοί έχουν να κάνουν με την επικουρικότητα. Ωστόσο, παρόλα αυτά, αν κοιτάξουμε στο παρελθόν τι έχει συμβεί στην πράξη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε κάποιες φορές συνδυασμός. Μέρη των μέτρων που θέλαμε να περάσουμε στην νομοθεσία ήταν κανονισμοί που υλοποιούνται αμέσως και μετά οδηγίε που πρέπει να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία. Αυτό εγκαταλείφθη βάσει της ε, λογικής της απλούστευσης, όμως η γενική εντύπωση που έχουμε αποκομίσει είναι ότι η απλούστευση έφερε πάρα πολλέ και πολύ δυσκίνητες μεγάλες οδηγίε, δύσκολες να μεταφερθούν και που απαιτούν να βρεθούν και συμβαστικές λύσεις οι οποίες δεν είναι πάντοτε εύκολο να εντοπιστούν. Και αυτές δυσχεραίνουν την μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας ε, ιδιαίτερος που ξεκινήσαμε αυτό το ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα. Ευχαριστώ λοιπόν και σας, ευχαριστώ, σας εύχομαι κάθε τύχη στις έρευνές σας και στο διακοπές των Χριστουγέννων, γιατί ξέρω ότι θα τις εκμεταλλευτείτε για να εργαστείτε και θα επανέλθουμε τον Ιανουάριο σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερος. Κλείνουμε την τελευταία μας συνεδρίαση για το 2010. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εδώ για τις μεγάλες τους προσπάθειες εκ μέρου. όλων μας επίσης ευχαριστίες προς το προσωπικό Τη επιτροπή μα και βεβαίω θα συνεργαστούμε με όλου του συζητητέ κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και να ευχαριστήσω το προσωπικό των ομάδων και τη Επιτροπή ξανά. Δεν θα συναντηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, αλλά ανεπισήμω τη Δευτέρα το βράδυ θα βρεθούμε στις 6.30 στο, στην αίθουσα C41 1 στην πλευρά κανάλι. Θα ετοιμάσουμε λοιπόν εκεί ό,τι χρειάζεται. Ο συνάδελφος ε, εδώ ετοιμάζει φωτογραφίες και εκθέσεις για να είμαστε απασχολημένοι και στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους εδώ για τη συμμετοχή σας. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, πολύ ωραίες διακοπές της πρωτοχρονιάς και με χαρά θα σας καλωσορίσω και τον Ιανουάριο για μια νέα χρονιά ενεργετική και γεμάτη δουλειά. Και πολύ φιλόδοξη. Να πω ότι πρέπει να αρχίσουμε την ε, συνεδρία των συντονιστών στις 11.30. Οπότε θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, γιατί ξέρω ότι ο κύριο Βάνιο πρέπει να φύγει.